I would like to uh, Θα σας την άδεια σας να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. ορίζοντας την Επίτροπο Μάλστρομ. Πριν όμως αρχίσουμε να συζητάμε την έκθεση PNR, κάποια θέματα στην ημερήσια διάταξη που θα ήθελα, να μου επιτρέπετε σύντομα, να σας εκθέσω. Σας ενημερώνω καταρχάς ότι η κυρία η εισηγείται και οι σκιώδεις εισηγητές συμφώνησαν την αναβολή της ψηφοφορίας ε, για την προτινόμενη οδηγία ως προς επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής που είχε αρχικά προβλεφθεί για αύριο. Αναβάλλεται λοιπόν και τα τέλη Μαρτίου κατόπιν αιτήματος της εισηγητρίας. Άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη μάλλον στι ανακοινώσει, είναι το εξή, ότι όπω ξέρετε έχουμε πολλή δουλειά στην ημερήσια διάταξη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματά μα, για αύριο η κυρία Γκέπχαρτ, η συγκήτρια για την γνωμοδότηση ω προ τα, καθεστώτα, τα γαμικά καθεστώτα και ο κύριος Μάικλ Κάσμαν, συγκητής ε, για τη γνωμοδότηση, τάξη γνωμοδότηση για τις συνέπειες της ε, κυριότητας σε καταγεγραμμένες, ε, αναγνωρισμένες σχέσεις ε, συμβίωσης, συμφώνησαν από κοινού να αναβληθεί η κοινή παρουσίαση των ε, γνωμοδοτήσεών τους για την 21η Μαρτυροχικά είχε προβλεφθεί για τις 28 Φεβρουαρίου. Επίσης, θα θέλω να σας αναφέρω ότι η κυρία Τιτ Πάουερ ορίστηκε πλήρες ε, τακτικό μέλος της Επιτροπής μας, ενώ ήταν μόλις αναπληρωματικό μέχρι πρόσφατα, την ορίζετε όμως όλοι πολύ καλά. Επίσης, Έχουμε τις εξής προτάσεις από την συνεδρία των συντονιστών για εισηγητές. Πολιετές πλαίσιο ε, για την ε, υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα η κυρία Ζανότκα για την περίοδο 2013-2017, ο κύριος Τρενταφυλλίδης για το άσυλο, ανταλλαγή, αρρωγή, εκπαιδευτικό σύστημα κατάρτισης ε, κυρία Μάκιντάιρ κατά της παραποίησης και αν δεν έχετε αντιρρήσεις εγκρίνω. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το λόγο ομιλώντας τη γλώσσα μου στο ουγγρικό και παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά ότι αισθάνομαι βαθύτατη οργή για το γεγονός ότι και τι ε, παρακολουθούμε με μεγάλη ε, προσοχή τα όσα λαμβάνουν χώρα στην Ουγγαρία και έχουμε μία πρόεδρο εδώ της ε, Επιτροπής, ε, την κυρία Γκέντς, η οποία ανέχθηκε τις ε, φρικαλαιότητες που επέτραψε, επέτρεψε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που, που οδήγησαν στο θάνατο πολλών πολιτών μας, συμπολιτών μας στην Ουγγαρία από πλευρά τη κυβέρνηση. Το γεγονό λοιπόν ότι έχουμε μια, πολιτική, Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία εξακολουθεί να βάλει κατά τη Ουγγαρία και παρόλα αυτά ανέχεται στο Προεδρείο, στη θέση του Προέδρου, την, ε, το πρόσωπο τη κυρία Γκιόντ, η Πρόεδρο διακάπτει την ομιλήτρια. Όχι, Πρόεδρε, έχω δικαίωμα στον ελεύθερο λόγο. Κυρία Μόρβη. Στην τελευταία συνεδρίαση, Πρόεδρε, συζητούσαμε ακριβώς το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. και ζήτησα από τον κύριο Μπουταχάζη το θέμα αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη. Έχει, ε, ζήτησα μάλλον να μπει το θέμα του κύριου Μπουταχάζη στην ημερήσια διάταξη. Έμεινε κρατούμενο πολιτικό επί τρία χρόνια ε, στι φυλακέ τη Ουγγαρία και αν του είχατε επιτρέψει να έρθει εδώ, αν του είχαν επιτρέψει να έρθει εδώ, θα μπορούσα να σα εξηγήσει τι δεινά περνάει στην Ουγγαρία. Αρχικά είχε γίνει δεκτή η πρόταση αυτή, στη συνέχεια όμως απερίφθη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εν τέλει ο κύριος Μπουταχάζη δεν ε, έγινε δεκτός ως προσκεκλημένος της ε, ε, συνεδρίασής μας. Πρώτον, δεν ήταν στην ημέρηση διάταξη. Δεύτερον, ήταν απόφαση των ομάδων. Σύντομη απάντηση και συνεχίζουμε με την ημέρηση διάταξη. Oh, yeah. No, I would like to ask, uh, θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Ταβάρες να κάνει μια στιγμή περίληψη των ε, διαπραγματεύσεων για τις ε, διαπραγματεύσεις σχετικές με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Ταβάρες. Ναι, Πρόεδρε, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, αν επισαρτάται σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών λέει ότι έχουμε αρκετά εκκρεμή ζητήματα να συζητήσουμε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω ότι έχουμε καταλήξει συμφωνία ως προς τα τρία κύρια ζητήματα. Ορατότητα της Βόρειας Αφρικής, ως μία από τις περιοχές που καλύπτονται από το περιφερειακό πρόγραμμα, από ένα περιφερειακό πρόγραμμα προστασίας που έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο και επιπλέον έγινε δεκτή και μια πολύ σοβαρή ε, προσθήκη το ζήτημα της, του απειλής της ζωής ή του κινδύνου, του κινδύνου βασανιστήριων για την επανεγκατάσταση. Ένα άλλο ζήτημα ήταν αυτό των υπηκών ε, του Ιράκ, που τώρα αντικαθίσταται ως έκφραση από την έκφραση ε, μεταναστών ή προσφύγων, μάλλον προερχομένων από το Ιράκ. Δηλαδή καλύπτονται και άλλες ε, υπηκότητες, όπως Φερρυπίν, Παλαιστίνη ή άλλοι. Στο άρθρο 80, η γνώμη του Κοινοβουλίου, άρθρο 80 της Συνθήκης, λέμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της ε, νομικής βάσης, γιατί λέμε ότι αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με την αλληλεγγύη και προς τους πρόσφυγες, αλλά και με την ε, εσωτερική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στην ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων κατάσταση, αλλά το Συμβούλιο δεν συμφωνεί. Και θεωρεί ότι είναι προβληματική η χρήση αυτού του άρθρου νομικής βάσης. Προτείνεται λοιπόν το άρθρο 80 να εισαχθεί ως αιτιολογική αναφορά ύστερα από τι διαβουλεύσει και έτσι το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο δεν είναι ικανοποιημένο γιατί δεν έγιναν διαβουλεύσει με το Συμβούλιο και έτσι με την ε, αναφορά του άρθρου αυτού, με την πίστη του άρθρου αυτό μέσα σε μια διολογική αναφορά, ενδέχεται να καταρρεύσει όλο το σύστημα. το 2014 δεν υπάρχουν ασφαλεί ορισμοί και γι' αυτό δεν θέλουμε να, έχουμε τους, ε, δεν θέλουμε να διατρέξουμε τον κίνδυνο αυτό και προτιμούμε να ζητήσουμε την ε, γνωμοδότηση τη Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων αλλά και τη νομική μα υπηρεσία, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για τροποποίηση νομική βάση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αποδεχόμενη την εισαγωγή με την πλήρη παραπομπή στο άρθρο 80 του κειμένου της ε, ε, αιτιολογικής αναφοράς που προτείνει το Συμβούλιο. Και όλα αυτά βέβαια εν ώψη και των συζητήσεων για την πολιτική στο νομικό πλαίσιο και τη επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική χρήση, την, ε, τη δυνατότητα αξιοποίηση του άρθρου 80 σε άλλε αντίστοιχε προτάσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα για τι τελευταίε εξελίξει, τι τελευταίε εβδομάδε. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ενδεχομένω να ολοκληρώσουμε την απόφαση αυτή σύντομα, στι επόμενε εβδομάδες. Ευχαριστώ. Έχουμε ζητήσει γνωμοδότηση λοιπόν ε, πραγματογνωμοσύνη από την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων για την υπόθεση αυτή. πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινωθεί στην ε, Σύνοδο Ολομελία τον Μάρτιο. Η ψηφοφορία για τη δεύτερη ανάγνωση σε επίπεδο τη Επιτροπή μα θα λάβει χώρα στι 21 Μαρτίου. Η τελική διέγκριση και ε, στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Μάρτιο στην, στις Βρυξέλλες, στην Σύνοδο Ολομελίας των Βρυξελών. Και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα για το οποίο είστε εδώ, το θέμα της ε, συμφωνίας ε, PNR μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε ότι έχει μακρύ ιστορικό αυτή η συμφωνία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Επίτροπο Μάλστρομ καταρχάς εδώ και τον Υπουργό των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας, κύριο Νικολάη Βάμεν, εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου που έχει που είναι εδώ παρόντες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και επίσης θα ήθελα να παρακαλούσω την κυρία Σόφι Νετφέλτ που είναι η συγγήτρια της έκθεσης αυτής να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Η Σοφία έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσία της Επιτρόπου όπως και εκπροσώπου του Προεδρείου δείχνει τη μεγάλη σημασία που δίδεται στο συγκεκριμένο θέμα. Ξεκινώντας με τα συμπεράσματα, θα λέω ότι όλοι είδατε την πρόταση έκθεσης που έκανα, που σας ζητώ να καταψηφίσετε ή να μην εγκρίνετε ακόμα, εν πάση περιπτώσει, την συμφωνία για τη μεταφορά των δεδομένων PNR, ατομικών στοιχείων επιβατών. Δεν μου αρέσει να σας προτείνω να απορρίψουμε τη συμφωνία, αλλά δυστυχώς είναι προφανές από τη διαδικασία την οποία είχα προτείνει εδώ και μία διετία ότι αυτό το οποίο ήθελα ήταν να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να υποστηρίξουμε όλοι. Αυτό ίσχυσε και στη συμφωνία με την Αυστραλία. Σε κάποιες φάσεις πρέπει να συμβιβαστούμε, δεν μπορούμε να έχουμε το 100% αυτών που επιθυμούμε. Καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία με την Αυστραλία, αλλά αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας τώρα δυστυχώς δεν είναι επαρκές σε καμία περίπτωση όσο και αν φανούμε φάνταστοι. Αν επανέλθει κανείς όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή το 2003, όταν ξεκινήσαμε δηλαδή τις διαπραγματεύσεις, θα διαπιστώσει ότι από τότε μετά από εννέα χρόνια διαπραγματεύσεων υπήρξαν τέσσερις μορφές της συμφωνίας αυτής 2004, 2007, 2009 και 2011. Η συμφωνία του 4 αμφισβητήθηκε, πήγαμε στο δικαστήριο, υπήρξε ακύρωση της τότε συμφωνίας, το πετύχαμε αυτό, όχι ακριβώς με τους όρους βέβαια τους οποίους εμείς είχαμε προτείνει, αλλά παρόλα αυτά. Εκείνη την εποχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε έτσι και εξουσία για να ψηφίζει για τις διεθνείς συμβάσεις. Αλλά παρόλα αυτά, αν το Κοινοβούλιο μπαίνει στη διαδικασία να αμφισβητήσει μια συμφωνία στο δικαστήριο, το κάναμε γιατί ε, θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει. Υπήρξε η ενδιάμεση συμφωνία του 2006, μετά η κανονική συμφωνία του 7, μετά από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας της Λισαβόνας μας ζητήθηκε να ψηφίσουμε εκ νέου, δεν ψηφίσαμε, γιατί είχα προτείνει σαν εισηγήτρια να αναβληθεί η ψηφοφορία και να ζητήσουμε την αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας συμφωνώντας να μην ψηφίσουμε θεωρεί κανείς ότι η συμφωνία του 2007 δεν ήταν καλή συμφωνία γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε δύο χρόνια να ψηφίσουμε απευθείας. Εμείς ορίσαμε τα κριτήρια για τη συμφωνία σε δύο ψηφίσματά μας το Μάιο και το Νοέμβριο του 2010. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες ακολουθούμε για να κρίνουμε την πρόταση τώρα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένου τομεί υπήρξε πρόοδος. Αλλά δεν νομίζω ότι η πρόοδος που συνετελέστη είναι επαρκής, δεν θεωρώ ότι είναι ουσιώδης και σίγουρα υπάρχουν και ορισμένα σημεία στα οποία τα πράγματα πήγαν πίσω. Υπάρχει θα έλεγα μια νομική υποχρέωση αν θέλετε στην Ευρώπη έτσι ώστε η χρήση των προσωπικών στοιχείων σε μια τέτοια θα έλεγα μαζική μάλιστα διάρκεια να ανταποκρίνεται σε ορισμένα κριτήρια. Ε, είχαμε θέσει το θέμα επανειλημμένα, δεν πήραμε απάντηση, δεν θα μας δοθεί απάντηση στα ερωτήματά μας αυτά, γι' αυτό πρέπει να περάσουμε στις λεπτομέρειες συμφωνίες. Πρώτον, περιορισμός των στόχων. Ο περιορισμός του στόχου ορίζεται στο άρθρο 4 και στις υπόλοιπες υποπαραγράφους. Η πρώτη υποπαράγραφος δίδει πράγματι μια σαφέστατα καθορισμένη μορφή περιορισμού των στόχων που μπορεί, για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συμφωνία αυτή. πολέμηση της τρομοκρατίας όπως το είχαμε ζητήσει και κατά πολέμηση του διεθνούς εγκλήματος σοβαρού διεθνού εγκλήματο. Οι νομικοί σίγουρα μπορεί να πούνε ότι ο ορισμό το 4-1... δεν είναι ο καλύτερο, αλλά μπορεί να σταθεί. Όμω υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Το 4-2... το 4-3 και το 4-4. Γιατί ενώ στο 4-1 λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τα δεδομένα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας, αν διαβάσει το 3 και 4 τότε σου λέει και για μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία μάλιστα δεν ορίζονται. Αν το αποφασίσει λέει ένας δικαστής, τι σημαίνει αυτό. Η αρχική διατύπωση ήταν ότι αν ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο. ο έλεγχος των φυσικών προσώπων στα σύνορα και ε, για άλλους λόγους. Τώρα δεν θα κάτσω να σας διαβάσω όλη την παράγραφο, αλλά αυτό λέει. Δυστυχώς λοιπόν τα άρθρα 4.2, 4.3 και 4.4 στην ουσία καταστρέφουν αυτά τα οποία προβλέπει το 4.1. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για έναν μεγάλο αριθμό στόχων που είναι εντελώς άσχετα με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διεθνούς εγκληματικότητας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε να είχαμε λύσει στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η περίοδος συγκράτησης των στοιχείων. Βασικά τα δεδομένα ε, θα κρατούνται χωρίς περιορισμούς, όχι 15 χρόνια όπως πιστεύουν ορισμένοι, αλλά χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Τα πρώτα 15 χρόνια ε, η πρόσβαση στα δεδομένα προοδευτικά θα περιορίζεται. Αυτό είναι καλό βέβαια, αλλά δεν είναι το ίδιο με την αφαίρεση των προσωπικών στοιχείων. Μετά τα 15 χρόνια τα δεδομένα θα είναι πλέον ανώνυμα, αλλά δεν λέγεται πώς θα γίνεται αυτό. Θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι η περίοδος συγκράτησης των στοιχείων δεν ορίζεται. Τα δεδομένα αυτά δεν καταστρέφονται. Αν πάτε τώρα στη συμφωνία του 2004, η περίοδος συγκράτησης των στοιχείων ήταν 2,5 χρόνια μετά από τα οποία καταστρέφονται τα δεδομένα. Και τότε είχαμε θεωρήσει ότι τα δυόμιση χρόνια ήταν υπερβολικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε τώρα μια περίοδο συγκράτηση των στοιχείων χωρίς περιορισμούς, αν και τα δεδομένα τα προσωπικά θα χάνονται μετά από τα 15 χρόνια. Κατά συνέπεια όπως είχαμε ορίσει και στο ψήφισμά μας του 2010 ότι δεχόμαστε μόνο το push, τη διαδικασία push προς τη ΣΥΠΑ και όχι τη διαδικασία pull από και το είχαμε ορίσει και στη συμφωνία επίσης με την Αυστραλία. Όχι push and pull λοιπόν, αλλά μόνο push. Κοιτάξτε, ακούω πάρα πολλές φωνές δεξιά-αριστερά και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, λέει η κυρία Ιντεβέλτ. Λοιπόν, η παρούσα συμφωνία επιτρέπει να υπάρχει το λεγόμενο pull, εκτός από ορισμένε περιπτώσεις με πολλές εξαιρέσεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν βρίσκω κανένα λόγο για να ισχύσει κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παίρνουν αυτό το οποίο θέλουν, θέλουν δηλαδή το push σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά pull. Σημαίνει ότι έχουν 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση στα δεδομένα. Οπότε έχουν όλα τα δεδομένα, τα έχουν όλα τα δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν login σε ευρωπαϊκά πληροφορικά συστήματα και δεν έχουν να το κάνουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ε, αγαπώ τους Αμερικανούς, εμπιστεύομαι τους Αμερικανούς, αλλά η εμπιστοσύνη είναι καλή, ο έλεγχος είναι καλύτερος και δεν δίνει κανείς δικαίωμα λογίν πρόσβασης σε τρίτες χώρες. Τώρα, δικαστική αποκατάσταση. Είναι προφανές ότι η αποκατάσταση δεν έχει, στον τομέα αυτό δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος από το 2004. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τα ίδια μέσα που έχουν οι Αμερικανοί πολίτες. Δεν έχουμε πλήρη μέσα στη διάθεσή μας. Η περαιτέρω μεταφορά στοιχείων δεν έχει βελτιωθεί, μπορεί να έχει βελτιωθεί λίγο η διατύπωση. Αλλά οι προϋποθέσεις παραμένουν ίδιες όπως και το 2004 και το 2007. Ευαίσθητα στοιχεία. Το 2004 η χρήση ευαίσθητων στοιχείων είχε απαγορευτεί πλήρως. Θυμάστε τη συμφωνία που είχαμε αμφισβητήσει στα δικαστήρια. Τώρα όμως επιτρέπεται κάτω από ορισμένες συνθήκες, οι οποίες δεν ορίζονται, επαναλαμβάνω. Δεν θα μιλήσω τώρα για την νομική βάση. Θα πρέπει να πούμε τώρα ποιες είναι οι συνέπειες του ναι και οι συνέπειες του όχι. Αν πούμε ναι, όπως το είχαμε κάνει σαν παράδειγμα στη συμφωνία SWIFT ή στη συμφωνία PNR με Αυστραλία. Τι θα συμβεί. Κανένας δεν είναι μάγος, αλλά νομίζω ότι κάποιος θα αμφισβητήσει τη συμφωνία αυτή στα δικαστήρια και οι πιθανότητες, οι δικαστές να μην εξετάσουν το πολιτικό πλαίσιο, αλλά να εξετάσουν το νομικό, αν θέλετε, υπόβαθρο της συμφωνίας, είναι θα έλεγα πάρα πολύ πιθανό. Είναι πολύ σαφές ότι οι δικαστές θα ελέγξουν το νόμιμο της συμφωνίας και όχι τις πολιτικές ευθύνες και συμφωνίες. Θα πρέπει εμείς όταν αποφασίζουμε κάτι να είμαστε βέβαιοι ότι είναι τεθωρακισμένο θα έλεγα σε επίπεδο δικαστικό γιατί αλλιώς θα αποδειχθούμε ανόητοι. Στο άλλο σενάριο, αν πούμε όχι, τι θα συμβεί αν πούμε όχι. Η πρόβλεψή μου είναι ότι τα δεδομένα θα συνεχίσουν να ρέουν. Δεν νομίζω ότι θα, σταματήσει, ή θα σταματήσουν οι υπερατλαντικές πτήσεις. Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις χώρες μέλη, τουλάχιστον όπως το έχουμε ελέγξει, έχουν διμερείς συμφωνίες υπογράψει με τη ΣΥΠΑ που παρέχουν τη νομική βάση για τη μεταφορά των δεδομένων είναι λίγο άκομψες συμφωνίες γιατί θα υπάρχουν 27 διμερείς αντί για μία πολυμερή. Αλλά υπάρχουν, νομικά πλαίσια υπάρχουν. Ένα πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει νομική βάση, τότε μπορεί να υφίστανται οι αερομεταφορείς πιθανότητες νομικής, αν θέλετε, λήψης δράσης εις βάρος τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι επαρκές όμως για να μας πείσει με το ζόρι να πούμε ναι στην προτινόμενη συμφωνία. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να γίνει περαιτέρω αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης. Όχι. Οι Αμερικανοί δεν έχουν πει σε καμία περίπτωση ότι θέλουν να αναδιαπραγματευτούν, ήταν από την αρχή ιδιαίτερα θα έλεγα διστακτικοί και να μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ζητούν πράγματα. Οι Αμερικανοί σαν κυρίαρχη χώρα έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν οδήποτε στοιχείο για οποιονδήποτε. Δεν μπορεί κανείς να τους το σταματήσει αυτό. Αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε είναι συγκεκριμένες εγγυήσεις έτσι ώστε να καλύπτονται νομικά οι μεταφορές αυτές των δεδομένων μια τελευταία παρατήρηση, την οποία δεν θα πρέπει να μειώσουμε τη σημασία της. Τι προηγούμενο δημιουργούμε. Υπάρχει μια εν λειτουργία συμφωνία με την Αυστραλία. Ψηφίσαμε και πετύχαμε ένα συμβιβασμό ο οποίος είναι αμοιβαία αποδεκτό. Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία η οποία διαπραγματευόμεθα. Συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση με τον Καναδά από το 2009 αν δεν κάνω λάθος. Από τότε τα στοιχεία μεταφέρονται στον Καναδά χωρίς καμία νομική βάση γιατί δεν υπάρχει η συμφωνία. Αυτό το λέω για αυτούς που πιστεύουν ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία θα σταματήσει η μεταφορά των στοιχείων. Όχι, δυστυχώς τα δεδομένα μεταφέρονται και χωρίς συμφωνίες. Και υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες ζητούν τη μεταφορά στοιχείων PNR. <clears throat> Τρεις χώρες ζήτησαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να διαπραγματευτεί. Μιλάμε για Κατάρ, Νότια Κορέα και Ιαπωνία. Άλλες χώρες είναι η Κούβα, η Νότιος Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ίσως και άλλες χώρες. Λοιπόν, είπαμε και τελειώνω εδώ, ότι όταν υιοθετήσαμε τη συμφωνία με την Αυστραλία, είπαμε ότι αυτό θα είναι το επίπεδο κατελάχιστον για τις περαιτέρω συμφωνίες PNR. Αν πράγματι είμαστε σοβαροί σε σχέση με ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι το 2004, δυνατότητα δηλαδή ε, πρόσβαση σε δικαστική αμφισβήτηση των μέτρων εις βάρος ε, συγκεκριμένων φυσικών προσώπων, η συμφωνία λοιπόν της Αυστραλίας είναι πρότυπο. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την προτινόμενη συμφωνία, κάτι το οποίο με λυπεί. Ευχαριστώ. πολύ. Η κυρία Πίτροπος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε προκειμένου να συμμετάσχετε σε τόσο σημαντική συζήτηση. Βρίσκομαι εδώ για να σας ζητήσω να συνενέσετε Τη συμφωνία για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι οι αρχές επιβολής νόμου χρειάζονται τα PNR για να ε, εξετάζουν τα θέματα. Δεύτερον, διότι αυτή η νέα συμφωνία αποτελεί μια σαφή βελτίωση της υφιστάμενης ε, συμφωνίας. Και τρίτον, διότι δεν βλέπω καμία εναλλακτική λύση που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των πολιτών. Για να το εξηγήσω πιο αναλυτικά και μετά να απαντήσω σε ερωτήσει, ε, να απαντήσω επίση και στα σχόλια τη ηγήτρια. Σχετικά με την ανάγκη χρήση το στο PNR, οι υπηρεσίε τη Κομισιόν ε, ε, έδωσαν στοιχεία επανειλημμένα στην Επιτροπή. Το σοβαρό διεθνέ έγκλημα και τρομοκρατία δημιουργεί μεγάλη ζημιά στι ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα στοιχεία PNR επιτρέπουν ε, την δίωξη παρόμοιων ε, εγκλημάτων και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου έγιναν τρομοκρατικές ε, έρευνες όπως το τρομοκρατική ενέργεια στο Μουμπάι, τον έκρηξη στο Τζιμπουλά και την έκρηξη στο Times Square. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα στοιχεία PNR. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε και συστήματα και προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε και ένα ευρωπαϊκό PNR. Δεύτερον, αυτή η συμφωνία, και θα ήθελα να πω από πλευρά μου, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο τη υφιστάμενη ε, συμφωνία του 2007. Αυτό ζητήσαμε από την Κομισιόν να διαπραγματευτεί το 2004 δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση διότι ήταν προσωρινή και είχε απορριφθεί από το δικαστήριο όχι λόγω περιεχομένου αλλά λόγω της νομικής βάσης. Ήταν εσφαλμένη, ήταν λάθος νομική βάση. Χάρη λοιπόν στην ευρεία συνένεση στο Συμβούλιο του Κομισιόν και το Κοινοβούλιο μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα το έγγραφο το οποίο ε, σε σχέση με το έγγραφο που σας παρουσίασα πέρσι το Μάιο κάναμε μια συλλογική εργασία ακούσαμε τις θέσεις ε, και των τριών θεσμικών οργάνων και ε, οθήσαμε τις ε, πολιτείες να δεχθούν και να κάνουν παραχωρήσεις. Αυτή η νέα συμφωνία είναι σαφής, υπάρχει, προσφέρει αμοιβαιότητα, προστατεύει τα στοιχεία, τα δεδομένα και καθιστά το σύστημα πιο αποτελεσματικό. Πολλές από τις βασικές ανησυχίες που εκφράσατε στο ψήφισμα του 2008 νομίζω ότι διασκεδάζονται γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα σημερινά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιωτικό βίο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Σε σχέση με την τρέχουσα συμφωνία είναι ένα ενιαίο κείμενο και ως εκ τούτου είναι νομικά δεσμευτικό περιλαμβάνει σαφούς ορισμούς σε ζητήματα όπως τρομοκρατία και σοβαρό διεθνές έγκλημα. Και αυτό δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου. Επίσης ε, ενισχύει και το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Η συμφωνία διευκρινίζει και περιορίζει τις δυνατότητες χρήσης ε, αυτών των δεδομένων από τις αρχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους τρομοκρατίας και για σοβαρό διεθνές έγκλημα ε, για ποινές που απαιτούν ε, φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, τριών ετών ηρκτή. Η συμφωνία περιορίζει την περίοδο διατήρησης των στοιχείων. Είναι η περίοδο κατά την οποία τα στοιχεία DNA μπορούν να αποθηκευτούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια περίοδο μέχρι 10 χρόνια για σοβαρό διεθνέ έγκλημα και μόνο για τρομοκρατικέ πράξει τα στοιχεία μπορούν να διατηρηθούν για 15 χρόνια. Και κάτι ακόμα διασφαλίζει ότι τα στοιχεία PNR αποπροσυμποποιούνται έξι μήνες μετά την διαβίβαση από τους αεροπορικές εταιρείε. Όσοι έχουν λοιπόν πρόσβαση αργότερα είναι πολύ περιορισμένος αριθμός προσώπων που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου. Οτιδήποτε, μετά πέρα αυτή την περίοδο, οτιδήποτε ε, προσωπικό θα διαγράφεται. Και Ό,τι σχετίζεται λοιπόν με ένα πρόσωπο διαγράφεται, καταστρέφεται με αυτή την προθεσμία. Υπάρχουν ε, διατάξεις ε, όπως αυτή που απαγορεύει την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων ε, και να μην μπορούν να κοινοποιηθούν στο κοινό μετά από κάποια ε, επίθεση στο διαδίκτυο. Ε, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων για προσωπικούς λόγους και το αίτημα για διαγραφή τους. Επίσης προβλέπει την προσφυγή σε ένδικα μέσα. η κοινή εξέταση στοιχείων μπορεί να εξετάζεται μόνο κατά περίπτωση αναφορικά με τη μέθοδο. Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη. Όλε οι αεροπορικέ εταιρείε θα πρέπει να μεταφέρουν στοιχεία μέσω τη μεθόδου push εντό διετία. Η ΆΤΑ μα διαβεβαίωσε ότι κάποιες εταιρείε που δεν μπορούν να εφαρμόσουν το push θα εξετάσουν το ζήτημα. Τα pool, η διαβίβαση pool θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη όπως ζητήσατε και θα αφορά μόνο έκτακτες ε, καταστάσεις. Αυτό δεν αναφέρεται στην Συμφωνία του 2007. Θα είναι περιορισμένη η χρήση από τις αρχές των ΙΠΑ και θα ελέγχεται από διάφορες ε, αρχές κάτι το οποίο ε, ενισχύει το θέμα της λογοδοσίας. Θα έχουμε κοινέ αναθεωρήσεις σε τακτική βάση και πλήρη αξιολόγηση μετά από τέσσερα χρόνια προκειμένου να εφαρμοστούν όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κρατούν σφραγισμένα τα, τους, τα αρχεία σε την, επίσης υπάρχουν ημερομηνίες για την ε, τερματισμό ή την ε, αναστολή εφαρμογής Αναγνωρίζω πως ε, μέλη της Επιτροπής σας ε, αλλά και του σώματος γενικότερα έχουν επιφυλάξεις και ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε μερικές από αυτές σήμερα, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Καμία διεθνή συμφωνία δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν δύο εταίροι που διαπραγματεύονται το συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, ε, παραχωρήσεων πάνω σε θέματα πολύ λεπτά για τις Πολιτείες. Και φτάνω στο τέλος της παρέμβασή μου. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, που είπε ότι περαιτέρω διαπραγματεύσει ε, με τι ΗΠΑ δεν είναι εναλλακτική λύση. Το Μάιο σα έβαλα ένα σχέδιο συμφωνία ε, μου είπατε πού θα επιθυμείτε να υπάρξουν βελτιώσει, κάποιε ενδείξει προέκυψαν και από το Συμβούλιο. Εργαστήκαμε σκληρά και αυτέ είναι οι τελικέ διαπραγματεύσει, οποίε καταλήξαμε πολλέ παραχωρήσει. Έγινε σίγουρα δεν είναι τέλεια η συμφωνία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο. Δεν υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα παραχωρήσεων από τι ΗΠΑ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς συμφωνία PNR, θα επηρεάσει τις διατρονικές μας σχέσεις, αλλά θα μας βάλει και σε μια κατάσταση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρείε ε, να διαβάζουν τα στοιχεία PNR και οι αεροπορικές εταιρείε θα το πράττουν. Και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη νομική αβεβαιότητα για τις ε, εταιρείε και επίσης οι πολίτες μας θα παραμείνουν χωρίς καμία νομική προστασία αναφορικά με το πόσο χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά στις πολιτείας και άλλες κράτη μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να επιβάλλουν τα ε, στοιχεία PNR στις πτήσεις τους και αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο ε, αν καταλήγαμε δεν θα είχαμε καμία δυνατότητα να προστατεύσουμε τους βάρη της Ένεσης. Για όλους τους λόγους λοιπόν κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Σα ζητώ να εγκρίνετε την ε, συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Βάμεν, πρόσωπο τη Προεδρία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου να ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, για την υποστήριξη των προσπαθειών μας. Η ισορροπία μεταξύ των αναγκών για τήρηση της τάξης, εφαρμογή του νόμου και το και την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών δεν ήταν ποτέ εύκολο έργο. Του Νοντήρου είναι πολύ πατητικό και σκληρό έργο και ήξερα πολύ ότι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα κάνει, επιτελεί το έργο της η Επιτροπή σας στην υπόθεση αυτή. Και γι' αυτό λόγο θεωρώ ότι η Προεδρία της Δανίας ε, είναι, ήταν σημαντικό να παρούσε εδώ για να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει ούτε μία αμφιβολία προς την τοποθέτηση του Συμβουλίου στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι δυνατό ποτέ να αναμένει κανεί σε μια διαπραγμάτευση ότι θα εξασφαλίσει όλα αυτά τα οποία προσδοκούσε όταν άρχισε τις διαπραγματεύσεις και αυτό ισχύει και στην ε, εν συμφωνία. Ε, βάσει και των οραμάτων που από κοινού είχαν ορίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διαπραγματεύσεων βάσει την εντολή που είχε για τη Συμφωνία PNR με τι ΗΠΑ. Ε, ταυτόχρονα ωστόσο ήταν πάντοτε σαφές ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας είχαν και αυτοί δικούς τους στόχους ορίσει. Στο σχέδιο λοιπόν ε, συμφωνίας πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ανάγνωση από αυτό το φως για να διαγνωστεί το πόσο σημαντικά επιτεύγματα έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία και συγχαίρω για τα καλά αποτελέσματα. Τούτου λεχθέντος δεν είναι τέλεια η συμφωνία που δεν είναι τέλεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν το τέλειο να, μετατραπεί, να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε εχθρό του καλού. Το σχέδιο έχει, καλή, έχει σημαντική προσθέμενη αξία για τον πολίτη. Προσφέρει ταυτόχρονα την ασφάλεια δικαίου που διεκδικούν, που ζητούν οι εταίροι μας. Έτσι λοιπόν, τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, επιδείξει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται και έχει με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσει το πιο σημαντικό, δηλαδή τα δικαιώματα των πολιτών μας και σημαντικό ρόλο για την συζήτηση τώρα ενός βελτιωμένου σχεδίου συμφωνία, στο οποίο χάρη προσπάθεια ακριβώ του Κοινοβουλίου μπορέσαμε να καταλήξουμε. Και επιτρέψτε μου λοιπόν εκ μέρου του Συμβουλίου τώρα να σα καλέσω να εγκρίνετε τη συμφωνία αυτή, να τη δεχθείτε. Δεν σα ζητώ να την ενστερνιστείτε. Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε και τι προσπάθειε ε, που ε, πραγματοποίησαν οι στενοί εταίροι μα, οι Αμερικανοί, για να ικανοποιήσουν τα δικά μα αιτήματα. Α ε, δεχθούμε λοιπόν τη συμφωνία αυτή ω τη βέλτιστη δυνατή καλή λύση Ας μην κοιτάμε τι δεν επιτύχαμε, ας κοιτάξουμε κυρίως αυτά που έχουμε επιτύχει. Και ε, με αυτό το πνεύμα ελπίζω το κοινοβουλίο σα να πει ναι στη συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ε, κύριε Γουάμεν, για, την, ε, για τις προτάσεις του Προεδρίου, του Συμβουλίου. Δεν ξέρω εάν η Σοφή Νετφέλτ θέλει να απαντήσει αμέσως. Μια διευκρίνηση μόνο, Πρόεδρε, όχι διδικαστικό. Προσπαθώ να καταλάβω το εξή, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ το Συμβούλιο να έχει ξαναέρθει να μας μιλήσει στο θέμα αυτό και να προσπαθεί να πείσει το Κοινοβούλιο να ψηφίσει προς μια κατεύθυνση. Το Συμβούλιο έχει ακολουθήσει τη δική του θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει τη δική του θέση. Όπως εμείς δεν πάμε στη συνεδριάση του Συμβουλίου να υποστηρίξουμε τις δικές μας τοποθετήσεις. Θα ήθελα να μου πει ο Πρόεδρος τι φρονεί για όλα αυτά, ο Προεδρεύων. Μπορούμε πιστεύω να αναβάλουμε προς το τέλος αυτή την απάντηση. Κύριε Νιθφέλτ, πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε θα παρακαλούσα η πρόεδρος ή ο πρόεδρος της Επιτροπής να μας δώσει γραπτή απάντηση προς τη διαδικασία. Θα μας απαντήσει ο κύριος Βάμελα ασφαλώς στο τέλος, αλλά... Ας δούμε πρώτα αυτού που θέλουν να λάβουν μέρος στη συζήτηση, καθώς είναι πολύ σημαντικό το θέμα και πρέπει να ακούσουμε τις απόψει των διαφόρων πολιτικών ομάδων πριν ε, δεχθούμε και τις απαντήσεις στα σχόλια αυτά. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα τους σκιώδεις συγκητές που έχουν στήσει το λόγο με τη σειρά και στη συνέχεια τους λοιπούς συναδέλφου, γιατί πολλοί άλλοι έχουν στήσει το λόγο. Κύριο Φού πρώτα, Σκιώδη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θα σας παρακαλέσω όσο το δυνατό να είσαστε σύντομοι γιατί περνάει ο χρόνος πολύ γοργά ως συνήθως. Ευχαριστώ καταρχάς. Είναι σαφές το πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε. Η κυρία Νετφέλτα έδωσε μια καλή ε, επισκόπηση της κατάστασης, ήταν καλό, ήταν κακό, ήταν επαρκές. Κανείς δεν θεωρεί μόνο ότι είναι τόσο καλή η συμφωνία που μπορούμε να αισθανόμαστε απόλυτη ικανοποίηση. Πολλά είναι τα προβλήματα, σαφές της πάση, Ωστόσο και εσωτερικά έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό όπως άλλωστε και την, προηγούμενη, την προπροηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο της Ολομιλίου Στρασβούργο με την Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Επιτροπής και με αίτημα προς την υπηρεσία προσωπικών δεδομένων ε, προς την οποία, από την οποία έχω λάβει απαντήσεις ε, που λένε ότι πρώτον έχει ελλείμματα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων της και τις σχετικέ προδιαγραφέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συμφωνία που όμως αποτελεί στην τωρινή μορφή μια σχετική βελτίωση. Δεύτερον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσαν να είναι χειρότερη θα μπορούσε να είναι χειρότερη εάν δεν υποστηρίζαμε αυτή τη συμφωνία για τους Ευρωπαίους πολίτες, λέει η απάντηση της Υπηρεσίας Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και αν κοιτάξουμε Άλλωστε και η κυρία Νετφέλτ στο σημείο 7 της εκθεσής, σας, το, της το έχει καταγράψει. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια περίοδο προσαρμογής, μια περίοδο ε, καταγραφής δεδομένων για τους πολίτε, των πολιτών την οποία θα μπορούσαμε να ελέγχουμε καθόλου ε, και εάν λαμβάναμε υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε τις εξελίξεις αυτές τότε ίσως η κατάσταση ε, η δικαιική κατάσταση που θα προξενούνταν από την απουσία συμφωνίας για τους πολίτες μας θα ήταν πολύ σοβαρή, πολύ κακή απαράδεκτη επίσης από πλευράς των ε, αεροπορικών εταιριών. και θα μπορούσε να τεθεί σε αμφιβολία από τις αεροπορικές εταιρείες ε, όχι μόνο η ισχύ της προηγούμενης συμφωνίας αλλά και η δυνατότητα η δικαιοπρακτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τέτοια διεθνή συμφωνία. Πράγματα τα οποία βέβαια πρέπει όλα να τα λάβουμε υπόψη και να τα σταθμίσουμε ως προς και βάσει αυτών των σταθμίσεων να καταλήξουμε σε μια πολιτική επιλογή και απόφαση. Μην ξεχνάμε δε ότι μπορεί να μιλάμε πάντα για τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους, αλλά έχει σημαντική ε, ε, παρουσία και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ασφαλώς η διάσταση της ασφάλειας στην υπόθεση αυτή. Η κατάσταση pull-push επίσης σημειώνεται εδώ πρόοδος πρέπει να πούμε και έτσι δεν είναι επαρκής και ικανοποιητική αλλά η μη τι άλλων ε, προς το παρόν ορίζεται ότι το pull, το pull δεν λαμβάνεται υπόψη ποτέ και στις ε, άκρους εξαιρετικές περιστάσεις. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα για μια ετήσια αναθεώρηση της συμφωνίας αυτής, πράγματα τα οποία εάν τα βάλουμε όλα κάτω και κάνουμε το λογαριασμό και τη σούμα, μας υποχρεώνουν πιστεύω να καταλήξουμε στο συμπέρασμα της έγκρισης της συμφωνίας, εφόσον θέλουμε να υποστηρίξουμε και να ε, εντείνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και ιδιαίτερως εάν θέλουμε να ε, υπάρχει η σωστή χρήση και αξιοποίηση των δεδομένων, γιατί έτσι βελτιώνεται η ασφάλεια δικαίου για όλους εμπλεκόμενους, έστω και αν η προτινόμενη συμφωνία δεν είναι η βέλτιστη. Καλώς λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Άλμπρεχτ επίσης και ο για την ομάδα του. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. οι θετικές, οι δυνάμει θετικέ αξιολογήσει και εκτιμήσει του προλαλήσαντο δεν με βρίσκουν ασήμαντο, πρέπει να πω. Εμεί έχουμε κάποιε επιφυλάξει που έχουν ήδη επισημανθεί από την εισηγήτρια, την κυρία Ενετφέλντ, έναντι αυτή τη ε, συμφωνία, τη προτινόμενη συμφωνία. Και το ερώτημα είναι ότι αν πρόκειται να ψηφίσουμε εδώ, ε, καταλήγουμε με την ψηφορία σε ένα αποτέλεσμα επιθυμητό, ναι ή όχι. Αυτό που βλέπω λοιπόν εδώ είναι ότι κάποια σημεία τα οποία διαρκώς επισημαίνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα όχι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, αλλά εδώ και 7-8 ε, χρόνια πλέον που έχουμε την υπόθεση αυτή μπροστά μας, είναι όλα τα σημεία στα οποία δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο, τα οποία θεωρούμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι προς τα αιτήματά μας και ιδιαίτερως δεν υπάρχουν σαφείς ε, ε, επιλογές, το profiling ότι δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει καθόλου σε σύγκληση, σε προσέγγιση. Το ζήτημα της σημαντικής μείωσης της περίοδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα ή το επίπεδο ε, δυνατότητας πρόσβασης, δηλαδή η κάλυψη μαζί με, το, με την περίοδο διακράτησης των δεδομένων για συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων μέχρι 10 έτη, οι Αμερικανοί μας λένε ότι όχι θα κρατάνε τα δεδομένα αυτά για όσο περίοδο, όσο περίοδο θέλουν απροσδιόριστη και η φύλαξη των δεδομένων αυτών, η επεξεργασία τους μπορεί να ε, οδηγήσει σε κάποια διαφορετική μεταχείριση μόνο εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να προκύψει παραβίαση των δικαιωμάτων. Δηλαδή είναι πολύ ασαφής η τοποθέτηση αυτή και έτσι εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχθούμε μία ε, διακράτηση των δεδομένων χωρίς ουδένα λόγο ή πρόσχημα που θα μπορούσε από έξι μήνες να φτάνει μέχρι και τα πέντε χρόνια και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εάν αναλογιστούμε πρώτα απ' όλα ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι ανοιχτή σε αρχές ε, χωρίς συμφωνία. Ότι δηλαδή μια τέτοια συμφωνία προσφέρει πολύ περιορισμένη βελτίωση ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων για, τη δική μας πλευρά τουλάχιστον, για δε την ασφάλεια δικαίως προς τις αεροπορικές εταιρείες. Για διαλογηθείτε, δηλαδή ότι μπορεί να έρθει μια η αδίποτε χώρα να τον κόσμο να έρθει και να απαιτήσει, ότι, να απαιτήσει τα τάδε τα δίνα προσωπικά δεδομένα από τις, από τις αεροπορικές εταιρείες και να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί σε αυτές τις απαιτήσει, πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει σε σοβαρές δυσκολίες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να δεχθούμε όλες αυτές τις πιέσεις και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να πούμε εμείς, να ορίσουμε εμείς ποια μέτρα θέλουμε, ποια μέτρα θεωρούμε θέμητα και ποια όχι. Και ιδάλλως θα ε, περιοριστούμε μόνο στην αποδοχή των μέτρων εκείνων που θεωρούμε ότι είναι αποδεκτά και θεμητά ως προς το δικό μας δικαιικό πλαίσιο. Το profiling, παραδείγματι, το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν βλέπω ότι θα πρέπει να υποχωρήσουμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δεχτούμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κέρκο, που επίσης είναι σκιώδης εισηγητής. Πρόεδρε, φτάνουμε σε μια κρίσιμη στιγμή τώρα δεν νομίζω ότι υπάρξει ένα άλλο θέμα το οποίο να έχει συζητηθεί τόσο πολύ από εισηγητές, σκιώδεις, συμβούλιο, επιτροπή, από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει, θα έλεγα, κάτι τέτοιο στο παρελθόν και όλοι όσοι προσπάθησαν θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι φτάσαμε σε μια στιγμή τουλάχιστον από μια πλευρά πολιτική πρέπει να ληφθεί απόφαση. Οφείλω να ομολογήσω ότι σέβομαι την εισηγήτρια και διαφωνώ με τα συμπεράσματά της. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια βελτιωμένη πρόταση μετά από τις συζητήσεις που είχαμε με την Επίτροπο μετά από τις συζητήσεις που είχαμε με το Συμβούλιο, μετά από τις χιλιάδες ε, συζητήσεις και τεκμήρια που πήραμε και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρώπη, είμαι πεπισμένος ότι πήγαμε καλά. Αν συγκρίνει κανείς αυτή τη συμφωνία με οποιασδήποτε άλλες έχουν υπάρξει, είναι καλή. Δεν μπορεί να πετύχουμε πάντα το 100% των ετοιμάτων μας. Αυτό δεν είναι δυνατόν στις διεθνείς συμφωνίες. Αυτό που έχει σημασία για μας όμως είναι ότι οφείλουμε εμείς να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης. Έχουμε την υποχρέωση να έχουμε ένα μέσο στη διάθεσή μας, σωστά ορισμένο, σωστά ελεγχόμενο, έτσι ώστε να μην διατρέξουμε τον κίνδυνο μιας αναρχικής διμερούς συμφωνία στην οποία δεν θα ελέγχουμε στο μέλλον, γιατί μια τέτοια συμφωνία δεν θα βοηθήσει στο μέλλον τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα στα πολύ ευαίσθητα θέματα και η πολιτική μου ομάδα θα υποστηρίξει την πρόταση αυτή. Έχει σημασία να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν εγώ δεν θα ήθελα να υπάρξει έλλειψη βεβαιότητας γιατί διακυβεύονται οι ζωές των πολιτών. Ξέρω ότι παθιαζόμαστε όταν συζητάμε τα θέματα αυτά, τις λεπτομέρειες, το 100% αυτών που θέλουμε να το αποκτήσουμε, αλλά ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Έναν κόσμο διαπραγμάτευσης όπου πετυχαίνουμε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε και νομίζω ότι πήγαμε καλύτερα από όσο ορισμένοι θεωρούσαν ότι πήγαμε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έκβαση. Έχει τις δικές της επιφυλάξεις η συγγήτρια, εγώ όμως θα στηρίξω την πρόταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τη Σοφή Ινβέλτ. Δεν συμφωνώ κι εγώ από τις εξελίξεις οι οποίες μας προτείνονται προς έγκριση. Δεν θα επαναλάβω όσα ακούστηκαν. Υπεψηφίζοντας μια τέτοια συμφωνία έχω την αίσθηση ότι εγκρίνουμε βήματα προς τα πίσω σε σχέση με τα δικαιώματα του πολίτη στην Ευρώπη. Δεν έχουμε καμία βεβαιότητα για την χρήση των στοιχείων αυτών στα άρθρα 12-13 σχετικά με τα δικαιώματά τους. Έχουμε να κάνουμε με μια δεδομένη πλέον νομική ανασφάλεια και στην ουσία δεν κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Αν υπεψηφίσουμε την πρόταση αυτή θα εγκρίνουμε αυτήν την νομική παλινοδία. Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από τους Αμερικανούς, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εφόσον δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι, πρέπει σώνει και καλά νομικά να εγκρίνουμε κάτι το οποίο μας πάει πίσω σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την οποία τόσο υπερηφανευόμεθα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πούμε ότι μιας και δεν πετύχαμε τίποτα περισσότερο πρέπει σών και καλά να εγκρίνουμε. Κυρία Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λαμβάνω το λόγο ξανά της ομάδας μου, μόνο ότι εγώ δεν είμαι σκιώδη συγγήτρια. είναι η κυρία Μπετζησί Πέλ που σήμερα δεν ε, μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίασή μας και μου ανέδεσε να εξηγήσω την θέση της ε, πάνω στην συμφωνία. Τώρα, οι γενικές γραμμές ε, της διαφωνίας ε, της κυρίας Χέπελ ε, ε, συμπίπτει με τα όσα ακούστηκαν όχι μόνο το πεδίο εφαρμογής που δεν είναι αναλογικό σε σχέση με τον επιθυμητό στόχο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διαβίβασης, παρουσία και χρήση του συστήματος pool μόλον ε, ε, είναι δυνατό σε έκτακτες περιπτώσεις ε, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό. Τώρα για την περίοδο διατήρησης, όπως είπε η συγγήτρια, μολονότι προκύπτει ανωνυμία των στοιχείων, τα στοιχεία όμως συνεχίζουν να υπάρχουν πάντα. Τώρα σε όλη φορά την θέμα της, των ένδικων μέσων και της προσφυγής δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επιτραπεί σε μια ουσιαστική προστασία. Μόνο ότι γίνεται ρητή αναφορά στην ε, διοικητική ή νομική δυνατότητα προσφυγής ε, στη ΣΥΠΑ, αλλά εδώ θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ε, θα μπορέσει να ευοδοθεί σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα με τις Αμερικανικές αρχές και δεν παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν την συμφωνία. Δεν αναφέρεται τίποτα το ρητό. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν η εισηγήτρια κυρία Σίπελ διαφωνεί με την συμφωνία να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία έκανε η κυρία Μάλστρομ αναφορικά με την προστασία των δεδομένων που εμένα μου δημιούργησαν κάποια σύγχυση. Θα ήθελα να γνωρίζω σε τι αναφέρονται η βελτίωση αναφορικά με, την, τα προσωπικά δεδομένα, επιθέσεις των κυβερνοχώρο, κάτι που είπε και το οποίο δεν κατάλαβα απολύτως. Ούτε εγώ ούτε ομάδα μου. Ευχαριστώ. Έξι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Κύριε Λάτφορπ, πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο θέμα της συμφωνίας αυτής είναι ότι δεν είναι απόλυτα ε, νομικά ορθό. Η νομική μας υπηρεσία το θεωρεί ότι εν μέρη είναι νομικά ορθό και αυτό συνδέεται με αυτό που είπε η συγγήτρια σχετικά με τα άρθρα 4.2, 4.3, 4.4. Φαίνεται, και ίσως αυτό να φανεί προκλητικό, ότι οι υπηρεσίε της Κομισιόν θεώρησαν πως αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε, ως εκ τούτου βασιζόμαστε σε μια επικοδομητική αμφιβολία. Θεωρούμε λοιπόν ότι με διαφορετικό τρόπο ερμηνεύουν οι δύο πλευρές, τα δύο μέρη την συμφωνία. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και διαφωνίες. Διότι δίνεται διαφορετική ερμηνεία όπου η πλευρά ισχυρίζεται ότι μόνο στα σύνορα μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 4 και 2 του 4-1. Νομίζω αυτό είναι ασφαλμένο και είναι κρίμα να καταλήξουμε σε αυτήν την ε, κατάσταση και θεωρώ ότι η συμφωνία δεν είναι κατάλληλη. Ευχαριστώ. Μια γενική παρατήρηση. Η συζήτηση που κάνουμε είναι πολύ σοβαρή. Γι' αυτό είναι η Επίτροπος εδώ, γι' αυτό είναι και ο εκπρόσωπος της Δανίας εκεί μπροστά σας και νομίζω ότι ναι μεν δεν έχουμε χρόνο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει στη δική μας Επίτροπη να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα ανάμεσά μας και να αποφασίσουμε ποια θα είναι η ψήφος επί τη βάση των συνεπειών αυτής της πιθανής ψήφου. Το να περιορίζεται το χρόνο συζήτησης σε αυτή τη φάση δεν είναι σωστό. Όλες οι εκθέσεις παρουσιάζουν ευαισθησίες και αντιθέσεις, αυτή επίσης και πολύ περισσότερο. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Δύο πράγματα όμως πρέπει να παραδεχθούμε. Πρώτον, χρειάζεται να προστατεύσουμε την ασφάλεια του πολίτη με πολλούς τρόπους. Ζούμε σε περίπλοκες εποχές και απαιτείται να κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάνουμε. Από την άλλη, είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτή τη συμφωνία, αν τη συγκρίνουμε με την προηγούμενη. Υπάρχουν επίσης και κάποια επιπλέον προβλήματα και θα πρέπει να ισορροπήσουμε τώρα τους σωστούς τρόπους λήψης απόφασης. Ταυτόχρονα θα ήθελα να κοιτάξουμε τις συνέπειες μιας θετικής ή αρνητικής ψήφου. Όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί από ό,τι φαίνεται εμείς είμαστε το τελευταίο όριο, είμαστε το τελικό όργανο αν θέλετε, το οποίο θα εγκρίνει ή μη μια διεθνή συμφωνία η οποία έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία χρόνια με άλλες συμφωνίες, το PFDP και πρέπει να πω ότι εγώ στα πλαίσια της πολιτικής μου ομάδας έδωσα μάχη για να υπεψηφιστεί η πρόταση αυτή η PFDP δεν είμαι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα και μιλάω για την δική μου πολιτική ομάδα, όλοι θεωρούμε ότι μας είχαν υποσχεθεί κάποια πράγματα και τελικά βλέπουμε ότι η χονδρική ε, μεταφορά δεδομένων συνεχίζεται. Και κάπου κάπου μας στέλνουν μία έκθεση γύρω από το πόσο καλά πάνε τα πράγματα και πόσο έχουμε βοηθήσει στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Πιο πρόσφατα είχαμε άλλο ένα παράδειγμα το οποίο δεν συνδέεται με την, με την Επίτροπο Μάστρομ για την άκτα. Αφού το διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή, αφού υπεγράφει από πάρα πολλά κράτη-μέλη, ξαφνικά βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη λένε «Επ, τι κάναμε εδώ» και δεν επικυρώνουν τη συμφωνία. Και φυσικά το βάρος πέφτει για μια ακόμη φορά για την άκτα σε μας. Και αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ακόμα και η Επιτροπή θέλει να προσφύγει στο δικαστήριο. Λοιπόν πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στους αερομεταφορείς, πόσο θα επηρεαστεί η ασφάλεια των συμπολιτών μας, ποιες θα είναι οι συνέπειες για την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μία τελευταία φράση. Ξέρω ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια ιστορία περίπλοκη. Και αυτό το ξέραμε εδώ και αρκετά χρόνια όταν συζητήσαμε το θέμα της απαλλαγής από, από βίζα. Γιατί κάθε φορά που υποχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε βάζουν περισσότερες απαιτήσει και ποτέ δεν δέχονται να κάνουν ένα βήμα το οποίο θα ωφελήσει και τον Ευρωπαίο πολίτη στο σύνολό του. Να πω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το θέμα αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό ακριβώς και παρατείναμε το χρόνο συζήτησης, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη μερίσια διάταξη και θέλω να δώσω το λόγο τώρα στους υπολείπους που ζήτησαν το λόγο να είναι πάρα πολύ ε, σύντομοι. Κοέλιο Μπουσούτιλ Γκόμες. Πρώτα όμως ο Ταβάρης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν δύο προβλήματα με τη συμφωνία αυτή. Το πρώτο είναι αυτό που ονομάζω οι δύο φάσεις και το άλλο που ονομάζω το άδωρο. Δηλαδή πρώτον, ε, στην ουσία κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός με το άρθρο 4, θετικό βήμα και μετά το καταστρέφουμε μέσα στο άρθρο 4. Με το 4-1 κάτι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε κάποιους περιορισμούς, πετυχαίνουμε κάποιους ορισμούς στην τρομοκρατική δραστηριότητα αλλά μετά στην ουσία ακυρώνουμε αυτό το βήμα το θετικό, επιτρέποντας στις άλλες παραγράφους τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και για άλλες ε, αφορμές και για το πώς θα χρησιμοποιούνται, πότε θα χρησιμοποιούνται, ε, με πολύ μεγάλο ποσοστό διακριτικής ερμηνείας από πλευράς της άλλης, ε, αν θέλετε, συμβαλόμενης πλευράς. Λοιπόν, ναι μεν έχει υπάρξει πρόοδος λοιπόν, αλλά με το δεύτερο βήμα αν θέλετε ακυρώνεται η πρόοδος αυτή. Δεν έχει νόημα μια τέτοια διαδικασία. Κάνουμε και ξεκάνουμε. Το άδωρο της υπόθεσης είναι η αποπροσωποποίηση των δεδομένων. Το έχω πει πολλά, πολλές φορές αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα αν αποπροσωποποιήσει κανείς τα δεδομένα και αντικαταστήσει το όνομα από μία σειρά από σύμβολα μετά από έξι μήνες, τρεις μήνες ή δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί έτσι και αλλιώ για ένα υπολογιστή είμαστε πάντα μία αλυσίδα συμβόλων και το όνομά μας είναι μία αλυσίδα συμβόλων. Πρέπει να υπάρξουν πολύ περισσότερες εγγυήσεις για το τι σημαίνει αποπροσωποποίηση. Θα πρέπει να συνδεθούν αυτού του είδους τα δεδομένα με το ανακτήσιμο σαν παράδειγμα του ονόματος ενός προσώπου. Δύο επιπλέον επιχειρήματα που ακούστηκαν. Πρώτον, ε, θα είναι χειρότερη η κατάσταση για τους επιβάτες αν πούμε όχι. Κοιτάξτε, θα έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια αν το θέλετε. Και η δυνατότητα αυτή θα ε, ισχύσει για να ενισχύσει τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δικαστικής αν θέλετε ζώνης. Δεύτερον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην είμαστε ασυνεπείς σε σχέση με το τι έχουμε πει ε, στο παρελθόν. Για να μας πάρουν σοβαρά πρέπει να είμαστε συμβατοί με τα επίπεδα τα οποία έχουμε ορίσει. Έχουμε πάρει αποφάσεις και πρέπει να τις σεβαστούμε. Μία τελευταία παρατήρηση. Η Βέμπερ έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να μην αγνοήσουμε τις προηγούμενες εμπειρίες. Με το SWIFT είχαμε πολλά προβλήματα εφαρμογής όταν ξεκινήσαμε. Είδαμε ότι οι εκθέσεις δεν μας έδιναν εγγυήσει για τη σωστή δίκαιη και αναλογική χρήση των δεδομένων SWIFT. Γιατί να μην μάθουμε από την εμπειρία αυτή παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία τώρα τι θα γίνει όμως με τα δεδομένα τα οποία έχουν ήδη στη διάθεσή τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λυπάμαι, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Κύριε Σκουέλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσω την τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε η Επίτροπος Μάλστον Θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσπάθεια που έκαναν σε διάφορους τομείς. Κάνατε μια καλή προσπάθεια. Η Επίτροπος Μάλστομ έχει δίκιο όταν λέγει ότι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις δεν πετυχαίνουμε ποτέ τα πάντα που επιθυμούμε. Το θέμα είναι αν το τελικό αποτέλεσμα είναι κοντά στο πρότυπο που θα θέλαμε εμείς να υπερισχύει στο πρότυπο το οποίο είχαμε προτείνει εμείς και το οποίο βασιζόταν στην Αυστραλιανή Συμφωνία. Υπήρχε πολιτική βάση, τα ε, ψηφίσματα του Τσολομέλειας και βέβαια συμφωνώ με πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασε η Σοφία Ιντεβελτ. Δεν μ' αρέσει η συμφωνία αυτή. Δεν μπορώ δυστυχώς να πω ότι είναι μια καλή συμφωνία Έχω σοβαρές αμφιβολίες για πάρα πολλά θέματα στα οποία ήδη αναφερθήκαμε. Αλλά υπάρχει εδώ ένα πολιτικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο τέθηκε και από την Σοφία Εντβέλτ, η οποία είπε ότι δεν φοβάται ότι αν τυχόν απορρίψουμε ε, την ε, συμφωνία ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Μας είπε η Εντβέλτ ότι η συνεχής ροή θα, θα παραμείνει συνεχής λόγω των διμερών συμφωνιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οπότε αυτό που μπορώ να πω στην εισηγήτριά μας για το συγκεκριμένο θέμα είναι ποιες είναι οι συνέπειες του όχι από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες στην ουσία ε, θα αντικαταστήσουν όλους τις άλλες διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στις Ένωση και τις τρίτες χώρες. Οπότε η κατάσταση δεν θα είναι χειρότερη. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο κύριος Μπουσουτήλ, έχετε ζητήσει το λόγο παρακαλώ γρήγορα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπό και την Προεδρία του Συμβουλίου που ήρθε εδώ. Συνήθως προσκαλούμε το Συμβούλιο να έρχεται εδώ για να παίρνει το λόγο. Τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Δεν συμφωνώ με τα συμπεράσματά της. Σέβομαι όμως, σαφώς, την προσπάθεια την οποία έκανε, ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο θέμα. Όλοι γνωρίζουμε, όπως είπε η Επιτροπή, ότι εδώ έχουμε μία συμφωνία ε, και ανεξαρτήτως του αν μας αρέσει ολόκληρη συμφωνία ή όχι, εδώ βρισκόμαστε. Και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ναι ή όχι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Ακόμα και αν υπάρχουν ορισμένα, εν πάση περιπτώσει, σημεία που μας αρέσουν και άλλα όχι. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τις συνέπειες των δράσεών μας αν πούμε ναι ή αν πούμε όχι. Στις ψηφοφορίες πολύ συχνά προσπάθησα να σκεφτώ τι θέλουν οι εκλογείς μου που με έστειλαν εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θέλουν είναι να μπορούν να πηγαίνουν στις Ηνωμένε Πολιτείες χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Αυτό που θέλουν είναι να μπορούν να πηγαίνουν στις Ηνωμένε Πολιτείες με ασφάλεια, δεν θέλει να τους τεινάξει κανείς στον αέρα, δεν θέλουν να πέσουν θύματα τρομοκρατικής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα θα συμφωνήσω ότι θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά χωρίς υπερβολική παρέμβαση στην προσωπική του ζωή. Και είναι αλήθεια ότι η συμφωνία αυτή δεν μας δίδει ότι εμείς θα θέλαμε, στα ψηφίσματά μας τα έχουμε άλλωστε εκφράσει. Και εδώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Κοέλιο να πω ότι Ακόμα και στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ένα θέμα είναι σαφές. Αν εμείς πούμε όχι στη συμφωνία αυτή, τότε οι συμπολίτε μας θα είναι σε χειρότερη θέση από ότι αν πούμε ναι. Και λέγοντας ναι σημαίνει ότι δεν θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε πετύχει ό,τι θα επιθυμούσαμε, είναι σαφές ότι αν πούμε όχι, τότε τα δικαιώματα των πολιτών μας θα αντιμετωπιστούν ακόμα χειρότερα. Κυρία Γκόμες, τελευταία ομιλήτρια. Ούτε μένα μου αρέσει η συμφωνία αυτή. Και νομίζω ότι και η πρόταση που είχαμε και πάνω στην οποία βασιστήκαμε, η Αυστραλιανή Συμφωνία, δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά. Και δεν πρόκειται για μια εκτελεστική συμφωνία για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έτσι και αλλιώς μπορεί να την αμφισβητούν συνεχώς το έχουν κάνει. Αυτό αμφισβητούν τις συμφωνίες σαν παράδειγμα την χρήση εδαφών στις χώρες μας, στις ε, στρατιωτικές βάσεις ας πούμε, που έχουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για δημοσιονομικούς λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν αμφισβητούν ότι έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο διεθνών συμφωνιών διμερών ή και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για δικαστική προσφυγή. Πέραν αυτού δεν έχω αμφιβολία ότι η απόρριψη σημαίνει ότι θα ισχύσουν οι εθνικές συμφωνίες οι οποίες δυστυχώς είναι χειρότερες. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω η συγκίτρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει η Σόφη ότι αυτό θα δημιουργήσει, αν πούμε όχι, σε ορισμένες δυσκολίες και εδώ και στη ΣΥΠΑ. Υπάρχει δυνατότητα το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθεωρήσουν την πρόταση αυτή και να διορθώσουν εκ των υστέρων έστω μετά την έγκριση ότι ότι ε, μας φαίνεται ότι δημιουργεί πρόβλημα. Κύριε Μάλστρομ, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας ε, και για την πολλή δουλειά που κάνατε. Μόνο ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στο τέλος. Άκουσα πολλές απόψεις, ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεργασία σας και Ακούσαμε ε, και οι θέσεις ε, του Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου πραγματικά ε, ήταν ικανοποιητικέ, συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά κλπ. Θα πρέπει όμως να δούμε το θέμα με ρεαλιστικό τρόπο. Τα κράτη-μέλη, τα κράτη μάλλον έχουν δικαίωμα να ζητούν στοιχεία για τους επιβάτες που εισέρχονται στο εδαφός τους και εμείς θέλουμε να το καταστήσουμε το δυνατόν ασφαλέστερο και σίγουρο για τους επιβάτες αλλά και να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου. Έχουμε λοιπόν ένα νομικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο που είναι ισορροπημένο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διμερείς ε, συμφωνίες είμαι πεπισμένη ότι η συμφωνία πληρεί αυτά τα που ζητήσαμε, όχι κατά 100% αλλά ε, έχουμε λάβει διασφαλίσεις ε, ικανοποιητικέ. Τώρα κάποιε διευκρινήσει για την περίοδο διατήρηση των δεδομένων. Είναι σαφέ ότι μετά από την αρχική περίοδο, σαν φέρετε στην ε, άρθρο 8, τα στοιχεία θα ε, και δεν θα υπάρχει δυνατότητα για μια επαναπροσωποποίηση των δεδομένων. Άρθρο 8.4 της συμφωνίας τώρα για την ασφάλεια των δεδομένων κυρία Ρομέρο Λόπες υπάρχουν επιπλέον διατάξεις πως αν υπάρξει κάποια επίθεση στον κυβερνοχώρο αυτά τα δεδομένα δεν θα επηρεαστούν. αναφέρονται στο διασυνοριακό έγκλημα το οποίο, για το οποίο προβλέπονται προβλέπεται κάθυρξη τριετής αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τώρα συγκρίσεις έχουν γίνει με την Αυστρία Χαίρομαι που τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν με τη συμφωνία αλλά η κατεύθυνση σαφής στην Επιτροπή σας, στο σώμα σας και σε όλες τις συζητήσει που είχαμε με εισηγητέ και εισηγητέ ότι η Αυστραλία από πλευρά Κομισιόν είναι το πρότυπο, το μοντέλο. Αλλά το Αμερικανική Συμφωνία θα είναι κατά διαφορετική. Για ποιο λόγο, διότι οι απειλέ είναι διαφορετικές από την Αυστραλία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν είναι ένα αντίγραφο της Αυστραλιανής Συμφωνίας, είναι μια συμφωνία την οποία επεξεργαστήκαμε ε, πολύ, λαμβάνοντας υπόψη ως βάση και την Αυστραλιανή Συμφωνία. Δεν συμφωνούμε λοιπόν σε όλα κατά 100% αλλά θεωρώ ότι πληρεί τις περισσότερες από τις ανησυχίες μας ε, ε, προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών μας, ε, την ασφάλειά τους ε, και θα μπορούσαμε να αλληλοσυγχαρούμε για την εργασία και το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Φυσικά μέχρι την τελευταία στιγμή της ψηφοφορίας οι υπηρεσίε μου και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριος Βάμεν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προκειμένου να μιλήσω ενώπιον σας, ε, χαίρομαι που είχα αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω την άποψη του Συμβουλίου στην Επιτροπή σας. Κατανοώ πως ε, η συγκήτρια και τα μέλη της ε, Επιτροπής σας έχουν αμφιβολίες και επιφυλάξεις για τη συμφωνία. Σέβομαι την άποψη αυτή. Η γνώμη της Προεδρίας ε, δεν ε, συμπίπτει με τη δική σας ε, ότι αυτή είναι μια συμφωνία την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία για να προσφέρουμε μια προστέμενη αξία στους πολίτες μας και όπως είπε και η Επίτροπος Μάστρομ υπάρχει κίνδυνος η απόρριψη της συμφωνίας να μας οδηγήσει σε ένα εναλλακτικό σενάριο πιο αβέβαιο και μη επιθυμητό. Πιστεύω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα, μπορούσαν, θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες εγγύσεις ε, προς όφελος των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ από την εισηγήτρια κυρία Ινβέλτ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Προτού να απαντήσω στα σχόλια θα ήθελα να κατηθήσω κάτι σαφές ε, για όλους όσοι παρακολουθούν τις συζητήσεις. Εάν καταψηφίσουμε τη συμφωνία και αν ε, δεν δώσουμε τη συμφωνία γνώμη, αυτό δεν σημαίνει ότι τα αεροπλάνα θα ανατινάζονται. Το 2010 στο ψήφισμά μας είχαμε πει ότι θεωρούμε ότι τα δεδομένα πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα. Αυτό το στήριξαν άπαντες στο σώμα το σώμα μας ποτέ δεν απέρριψε την χρήση προσωπικών δεδομένων για λόγους ασφάλειας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές ε, οι ιστορίες εκφοβισμού δεν έχουν ε, χώρο ύπαρξης ε, στην σημερινή μας συζήτηση. Δεύτερον, συνάδελφοι, ο διάβολάκος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και αν ακούμε πάντα γενικές συζητήσεις ότι η συμφωνία περιέχει ορθές λύτρες για την προσέγγιση δεδομένων και ε, ε, απαραίτητες νομικές προστασίες κλπ. Αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε όλοι το κείμενο. Σας καλώ. Ο διάβολος λοιπόν βρίσκεται στις λεπτομέρειες, διότι ειλικρινά ελάχιστες από τις αμφιβολίες μου και τις φυλάξεις που εξέφρασα αρχικά απαντήθηκαν από την Κομισιόν. Τώρα για τον ε, περιορισμούς ε, όλοι θεωρούμε ότι τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τρομοκρατία ή την καταπολέμηση του διεθνού εγκλήματος. Αλλά αποκλείουμε άλλε περιπτώσεις όπως τελωνία, ε, μεταναστευτικού ελέγχους και δημόσια υγεία. Δεν έχουν καμία σχέση με την ανατείναξη αεροσκαφών. Συνάδελφοι, σκεφτείτε πως τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξε μαζική συλλογή δεδομένων, μαζική και ποτέ δεν ε, οδήγησε αυτό σε πρόληψη τρομοκρατικών πράξεων. Ακόμα και ε, την 10η Σεπτεμβρίου οι μυστικές υπηρεσίες είχαν τα, τους τρομοκράτες στα ραντάρ τους. Λοιπόν, ας μην ε, ισχυριζόμαστε ότι η μαζική συλλογή δεδομένων θα θα μπορέσει να προλάβει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Και επίτροπε, η συμφωνία και αν διαβάσετε τα εναξιολόγηση του Ευρωπαίου Επόπτη Δεδομένων θα δείτε ότι και αυτό συμφωνεί με μας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ε, ε, αφησημίες. Ε, δεν μας ζητήθηκε να βρούμε λύση, μας ζητήθηκε να ε, στηρίξουμε ένα συμβασμό, διότι ναι, όντω ζούμε στον πραγματικό κόσμο, αλλά πρέπει να, είναι σύμβατη αυτή η συμφωνία με την Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Όνεσης Και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορώ λοιπόν να το συμφιλιώσω με την ε, συνείδησή μου και με τη σκέψη μου το γεγονός ότι θα ε, συμφωνήσω με μια συμφωνία η οποία ε, αντιβαίνει του ενωσιακού δικαίου. Ε, ε, προτείνω να συντομεύσω, διαφορετικά θα ξενυχτήσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την συμφωνία του 2004. Ήταν, δεν ήταν προσωρινή συμφωνία, ήταν μόνιμη. Απλά κατέστη προσωρινή διότι απορρίφθηκε από το δικαστήριο για λόγους διαδικαστικούς, διότι το δικαστήριο δεν τόλμησε να μπει στην ουσία. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισχυριζόμαστε ότι το 2004 υπήρχε μία απλή γνωμοδότηση. Η Επίτροπος ε, είπε ότι αυτή η συμφωνία διευκρινίζει αλλά και περιορίζει τον στόχο. Εγώ δεν θέλω να το διευκρινίζει, θέλω να τον περιορίζει. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος Ταβάρες, περιορίζει τον στόχο του άρθρου 4.1 και μετά όμως διευρύνει τον στόχο στο 4.2, 4.3 και 4.4. Ε, λέγεται ότι επιβολή νόμου αφορά την ε, απειλή στι ΗΠΑ. Κοιτάξτε, αν ε, εμεί πρέπει να υπογράψουμε μια συμφωνία, εμεί πρέπει να φροντίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας, πρωτίστως. Νομίζω ότι τα άπα σχετικά με το push pull, το ε, υποχρεωτικό για τους αερομεταφορείς να, μετα, μεταφερθούν στο ΠΟΥΣ μετά από δύο χρόνια. Με αυτό ήταν ο σκοπός και από το 2004. Ξέρουμε ότι αυτή η υποχρέωση δεν μπορεί να επιβληθεί. Εσύ το, κάτι το οποίο λέτε δεν ε, μπορεί να επιβληθεί μόνο από τις αρχές επιβολής του νόμου που θα επιβάλλουν κάποια πρόστιμα μερικών χιλιάδων ε, ευρώ. Αλλά σκεφτείτε και την επένδυση που θα κάνουν οι αερομεταφορείς για να μεταφερθούν το ΠΟΥΣ στο πουλ. Κοιτάξτε συνάδελφοι, εδώ δημιουργούμε προηγούμενο. Οι επόμενε χώρε που θα χτυπήσουν την πόρτα μα ενδέχεται να είναι η Ρωσία και η Κίνα. Τι θα πούμε. Θέλουμε δεδομένα σύμφωνα με, ε, με τη συμφωνία με τι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με την Αυστραλία. Η Κίνα θα το θέλει αυτό. Και εμείς θα πούμε δεν θέλουμε να σα τα παρέχουμε μας υπενθυμίσουν ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την ε, Κίνα να μας ε, διασώσει από την οικονομική κρίση. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τώρα τη σωστή λύση και όχι στο μέλλον σε ενδεχόμενες συμφωνίες με άλλες χώρες. Τώρα, το, ε, η συμφωνία αυτή είναι καλύτερη από μη συμφωνία. Όχι, δεν συμφωνώ διότι επαντλημένα ζητήσαμε όλους τους ε, νομικούς εμπειρογνώμονες και την Κομισιόν να μας πει τι διασφαλίσεις έχουν με αυτή τη συμφωνία οι πολίτες παρά με μη συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Η συμφωνία λέει ρητά ότι δεν μπορεί να προκύψουν δικαιώματα από την εν λόγω συμφωνία για φυσικά οι νομικά πρόσωπα. Δεν μπορούν να ε, προκύψουν. Η μόνη προστέμενη αξία της συμφωνίας αυτής είναι ότι προβλέπει ε, ασφάλεια δικαίου στους αερομεταφορείς. Ναι, είναι ορθό αυτό, είναι σωστό, κάτι με το οποίο συμφωνώ. Αλλά το πρόβλημα είναι η μοναδική προστέμενη αξία της συμφωνίας. Είναι ικανός λόγος λοιπόν προκειμένου να υπογράψουν μια συμφωνία που δεν είναι με τον, με το ενωσιακό δίκαιο και δεν προστατεύει τους πολίτες μας ε, περαιτέρω. Ε, μας, μας ζητείτε εδώ να νομιμοποιήσουμε κάτι το παράνομο. Και κατά λίγο Πρόεδρε, θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό κάτι το οποίο υπογραμμίζει και η παρουσία της Επιτρόπου και του εκπροσώπου της Προεδρίας. Και ένα τελικό σημείο σχετικά με τις αναθεωρήσεις. Έχοντας την δυνατότητα της αναθεώρησης, εντάξει μπορείτε να αναθεωρήσετε μια κακή συμφωνία αλλά παραμένει κακή η Ρενάντε Βέμπερ και εγώ, βλέποντας την εμπειρία που είχαμε με το SWIFT, έχουμε ελάχιστη εμπιστοσύνη σε μια κοινή αναθεώρηση. Και αυτοί που αναλαμβάνουν την ε, αναθεώρηση δεσμεύονται από ε, τον απόρριτο τον εμπιστευτικό χαρακτήρα. Παρακαλώ, μισό λεπτό, Πρόεδρε ακούσαμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ζήτημα. Οι κοινέ αναθεωρήσει του παρελθόντος αποκαλύπτουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για λόγους πέραν αυτών που είχαν συμφωνηθεί. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να εμπιστευτώ πω οι μελλοντικέ ε, αναθεωρήσεις, κοινέ αναθεωρήσει θα είναι καλύτερε. Κατανοώ πως αν καταψηφίσουμε θα βρεθούμε σε μια προβληματική κατάσταση. δεν είναι καταστροφή, θα είναι καταστροφική, αλλά προβληματική. Προσπάθησα να καταλήξω αποτέλεσμα που θα είναι καλύτερο. Δύο χρόνια το προσπαθούμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ως εισηγητρία πριν από δύο χρόνια, συνέθεσα στο σώμα μας να ε, σταματήσουμε τις ψηφοφορίες και να προωθήσουμε να αναδιαπραγματευτούμε. Αυτό το είχα προτείνει ω ε, συγκίτρια Προδιατία. Λυπάμαι λοιπόν ε, μετά από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων με του στενούς μα φίλου και ε, συμμάχους δεν καταλήξαμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και λυπάμαι που δεν μπορώ να συστήσω στο σώμα να, να υποστηρίξει τη συμφωνία. Πρόεδρο, ε, να διακόψουμε εδώ τη συζήτηση, θα ψηφίσουμε στι 26 Μαρτίου. Έχουμε λίγο χρόνο λοιπόν στη διάθεσή μα. 26. 26. 26 είναι κυρία Νατφέλτ. Θα επιβεβαιωθεί εδώ μεταξύ βέβαια. Μπορούμε να συζητήσουμε για τι τελευταίες λεπτομέρειες. ευχαριστώ θερμά. Έχουμε πολλά ακόμη ακριβή ζητήματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες του να εγκρίνουμε η μη τη σύμφωνη γνώμη μεταξύ μα. Σα ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σα. Okay, uh, go back to our seats, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξανακαθίσουμε σας παρακαλώ θερμά. Εξαιτία μου αρχίζουμε τώρα και καθυστερούμε, χάνουμε, ε, έχουμε καθυστέρηση στο πρόγραμμά μας. Άρα θα επιταχύνουμε τώρα. Αυτά έχουν. Ο πρόεδρος έχει αυτά τα προνόμια. Τώρα έχουμε την ημερήσια διάσταση, την ημερήσια διάταξη παρουσία από τον κύριο Μαρτίνου, ο οποίος είναι υπεύθυνο ε, για τα θέματα διακυβέρνηση της Europol. Θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα 2012 με μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, Πού είναι τα γυαλιά μου. έρχεται, άρα μπορώ να μιλάω ακόμα. Να φάμε χρόνο λίγο. Ε, συζήτηση που είχαμε το 2011 στην Επιτροπή μας. Και σα, μια και ήρθετε το μεταξύ σας δίνω το λόγο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με εσά για να λάβουμε το λόγο οι συνάδελφοι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Στο συγγνώμη που καθυστέρησα. Είναι ο κύριος Μαρτίνου. Καλησπέρα σας. Ο διευθυντής μας, ερχόμενος εδώ, κύριος Wainwright, είχε ένα ατύχημα το αυτοκίνητό του, ένα πρόβλημα μάλλον, έμεινε η μηχανή, από μηχανή και έτσι έστειλε εμένα άρον άρον ως αναπληρωτή διευθυντή. Εγώ έχω πρόσφατα ενταχθεί στους κόλπους της Γεωργοπόλη μόνο τον Νοέμβριο. Είμαι υπεύθυνο διακυβέρνησης, διοίκησης, οργάνωσης. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη μου επίσκεψη εδώ στο κοινοβόλιο γιατί ως ε, αρχηγός της αστυνομίας στη χώρα μου, ήμουν ε, αρκετές φορές προσκεκλημένος στο κοινοβούλιο, όμως ως εκπρόσωπος της Europol πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Το πρόγραμμα λοιπόν της Europol για το 2012 θα σας παρουσιάσω και ξεκινώ με στοιχεία από τις προσφατές επιχειρησιακές δραστηριότητες της ε, Europol και στο πλαίσιο του προγράμματος του 2012 ε, από τις αρχές δηλαδή, του έτους. Και παραδείγματα όπως ε, δίμευση 100 κιλών αμφεταμίνης, σημαντικές, ε, σημαντικών ποσοτήτων προδρόμων ουσιών, ε, εξοπλισμού, όπλων, πυροβόλων σε διάφορα κράτη-μέλη σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση μαζί με αυτή η οποία έβαινε κατά της παραγωγής, ε, ε, λαθρέας παραγωγής ναρκωτικών στους δρόμους. Ε, παράλληλα λοιπόν Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, κατοχώρες διελήθη ένα μεγάλο δίκτυο και παραγωγής και διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών ασφαλιστικών ουσιών. Πλην όμως ε, χωρίς να είναι η πιο σημαντική ήταν η τελευταία αυτή η επιχείρηση κοινή δράσης ταυτόχρονης για την καταπολέμηση του εγκλήματο και των ναρκωτικών και της κρίσης αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύει την ε, μεγάλη σημασία, τις ε, μεγάλες και ισχυρές υποσχέσεις και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και με την υποστήριξή μας, την υποστήριξή σας για την, υποστήρι... την ανάπτυξη του δυναμικού μας, των ε, τεχνολογικών μας δυνατοτήτων και του λογισμικού μας τώρα, του, της επιμελητίας μας μάλλον, αν μου επιτρέπετε τώρα θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την στρατηγική μας στρατηγική. Η πενταετής λοιπόν 2010-2014 προβλέπει ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμο για την ε, ανάπτυξη του δυναμικού ως ένα πρωτογενές κέντρο ε, στήριξης για τις διασυνοριακές ε, δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφύλαξη, εξασφάλιση πληροφοριών και κέντρο περιαγωγής των πληροφοριών αυτών επίσης οι ευθύνε μα, αναπτύσσονται μέσα από το τελικό κανονισμό με, το σχέδιο, με την απόφαση για τη θέσπιση τη Europol και σημαίνουν έκφραση των στρατηγικών φιλοδοξιών μέσα από ετήσιες ε, προγραμματικέ δηλώσει και οργάνωση τη υπηρεσία μα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό έχουμε σημαντικέ και εκτεταμένες εξωτερικέ διαβουλεύσεις με τι αρχέ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Europol και λοιπόν υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Στο πρόγραμμα δράσης Europol επίσης προβλέπει νέες εξελίξεις ως προς τη χάραξη πολιτικής και αξιοποίηση των μέσων που έχει έτσι ώστε να είναι πιο ουσιαστική η λειτουργία της υπηρεσίας τι μπορεί να επηρεάζει τώρα τους στόχους του 2011. Η συνθήκη της Λισαβόνας πρώτα απ' όλα, όπου η Europol ε, υποχρεώται να λογοδοτήσει σε μια ευρύτατη ε, γκάμα εμπλεκομένων φορέων. Ε, τώρα ζητούμε να βελτιωθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών και στα μέλη του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μας ζητείτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες και έτσι θα αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε για να ε, συνεργαζόμαστε και πιο στεχνά, ιδιαίτερα από το 2012. Επίσης, η απόφαση του Συμβουλίου για την Europol προσφέρει βάση και νέες ευκαιρίες βελτίωσης των υπηρεσιών προσφέρει η Europol. Φέρει πίν συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και διάταξη που επιτρέπει στη Europol να αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες και κοινέ ομάδες ερευνών Η απόφαση του 2011, όπως έχει εγγραφεί μέσα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011 και διάφοροι κύκλοι ευρωπαϊκής πολιτικής ορίζουν επίσης ε, δραστηριότητες και ύστερα από τις επιθέσεις στην Νορβηγία τον Ιούλιο του 2011 η Europol έχει δεσμευτεί επίσης να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2012 που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν ε, την VA τις βίαιες ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις ε, και ιδεολογίες και επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα διαλειτουργικότητας ε, όπου σε παιδό Europol επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα για ένα κοινό πρόγραμμα, ε, μάλλον πλαίσιο δράση για ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Αυτοί είναι οι παράγοντε βάσει των οποίων κινούμαστε μαζί με τη στρατηγική της ε, Europol που αποτελούν και τη βάση για, τις, ε, για τους 23 στόχους προτεραιότητας ε, που έχουμε ορίσει το πρόγραμμα το 2012. Και τώρα, αν επιτρέψετε, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιου από τους στόχους αυτούς. Η Europol θα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος δράσεως για το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα ευθύνη και υπευθυνότητα για την ανάπτυξη των διαδικασιών αυτών εφέτος συνεπάγονται ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας για αξιολόγηση του σοβαρού οργανωμένου κλίματος του 2013 αναμένεται να κατατεθεί με στόχο να προσφέρει σαφή και διαφανή μεθοδολογία Στηριζόμενη σε μια ποιοτική ανάλυση των κινδύνων συμπεριλαμβανομένων και λαμβανομένων υπόψη μια σειρά παραγόντων και όχι μόνο της επιβολής του νόμου. Επίσης, στήριξη στα κύρια κράτη για την εφαρμογή των ε, δράσεων λειτουργίας του 2012 και τρίτον διευκολύνουμε την προσοχή γύρω ε, της ε, λειτουργίας το 2013 και μετά με πολιτική δράση το 2013 με το όνομα ΑΕΡΕΑΣ, δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε στο δυνατόν πιο σημαντικές ε, τάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσουμε την μοναδική επισκόπηση που έχουμε των ε, υπερσυνοριακών ε, εγκληματικών δραστηριοτήτων. Θα βοηθήσουμε τις ε, χώρες μέρη να, στον εντοπισμό των χώρων εγκληματικότητας που μπορεί να αναπτύσσονται με βάση ένα δίκτυο διαθέσιμο ανα πάσα στιγμή σε 24 ώρη βάση και προσφέρει παρακολούθηση υποπτία και με αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων ε, εξοπλισμού παρακολούθησης και επικοινωνίας που έχουμε στα νέα μας κτίρια. μάλλον ε, λειτουργική στήριξη είχαμε και σε επίπεδο κλιματολογικό και ανάλυσης ε, και υποστήριξης με στόχο να στηρίξουμε και να ολοκληρώσουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ερευνών, ποιότητα δηλαδή και ποσότητα για μια νέα ανάλυση της δουλειάς αυτής που θα παρουσιάσει το 2012. Κοινό, εποπτικό όργανο, γραφείο προστασίας δεδομένων που συνεργάζονται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της AWF, ε, το νέο πλαίσιο δηλαδή, που θα μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε ανάλυση διασταύρωση πληροφοριών με βάση το εφιστάμενο AWF, να βελτιώσουμε τις ε, αναλύσεις τάσεων και τη διερεύνηση πιθανολογούμενων τάσεων σε δραστηριότητες εγκληματικές αλλά και παράνομα έσοδα που προκύπτουν από την ε, από τη λαθρομετανάστευση, το χείρισμα των θρομεταναστών, τα ναρκωτικά και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Πρέπει να πούμε επίση ότι το διαδικτυακό έγκλημα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μια έκθεση και μεγαλύτερη υπηρεσία ασφάλειας, στον, ε, στον ηλεκτρονικό χώρο μας έλεγε ότι ήταν πάνω από 290 δισεκατομμύρια οι απώλειες σε έσοδες Ε, πάνω από 290 δισεκατομμύρια λοιπόν ευρώ απώλεια εισοδημάτων, αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότηση ε, εγκλήματος οργανωμένου που έχει να κάνει ε, με το δραστηριότητες, μεταξύ των ναρκωτικά και τα όπλα. Η Εύρωπολ λοιπόν στην υπόθεση αυτή μπορεί να προσφέρει ενισχυμένε δυνατότητε για τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του ε, ε ανά τι χώρε με έναν τρόπο οργανωμένο, ολιστικό, πάλι μέσα από το πλαίσιο AWF και επίσης θα, θα αντιμετωπίσουμε και άλλες παράλληλες ε, μορφές εγκληματικότητας όπως παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Θα έχουμε συνεργασία με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες ΕΝΕΣΑ και Eurojust και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αντίσταση την εσωτερική στο ε, κυβερνό έγκλημα. Επίσης, Προσπαθούμε να συνεργαστούμε επιτυχώς και με τις, ετε... με τις ε, υπηρεσίες εταίρους, παράλληλες υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω και από αυτήν. Το 2012 θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις... Ε, τη συνεργασία μας και με τις υπηρεσίες εσωτερικών ε, και δικαιοσύνης αλλά και ταυτόχρονα με άλλους παράγοντες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιντερπολ, Ηνωμένες Πολιτείες, υποψήφιε χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες ε, μέσα από διάφορα προγράμματα όπω το ΜΑΟ και το ΣΥΚΛΑΤ. Για τις δραστηριότητε του οργανωμένου εγκλήματος ε, που βρίσκονται εκτό των κυρίων τομείων προτεραιοτήτων τώρα θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε ε, την πρόβλεψη εσωτερικών κινδύνων με πρόωρο σύστημα προειδοποίησης. Όταν ε, μπορέσουμε λοιπόν, για να ενισχύσουμε μάλλον τις τεχνικές δυνατότητες και τη διαχειριστική, το διαχειριστικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής, ε, ε της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Europol, είναι, έχουμε το σύστημα CNR, που είναι ένα σύστημα πληροφοριών, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Europol κρατών μελών και τρίτων κρατών, το οποίο θα εισαχθεί μέσα σε, θα ενσωματωθεί στα εθνικά συστήματα στα κράτη-μέλη και έτσι θα επιτρέψει στη Europol να συμμετέχει περισσότερο εκ του σύνολου και στις, ε, στις έρευνες ανά την Ευρώπη. Ταυτόχρονα εφέτος θα αναπτύξουμε και ένα ε, help desk, μια θηρίδα δηλαδή στήριξη των κρατών μελών ως προς την πρωτογενή εφαρμογή του συστήματος ε, για την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Επίσης, η Europol αναπτύσσει την ε, ανταποκρισιμότητά της στις ε, ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμβάθυνση στην ε, ανταπόκριση της προσδοκίας και ανάγκες των κρατών μελών και των ερευνητικών αρχών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε αλλαγέ. Έχουμε λοιπόν νέα καθήκοντα και σημαντική ε, ζήτηση για τις υπηρεσίες μας σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Ε, οι πόροι είναι περιορισμένοι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων μας και θα χαρακτηρίσει πιστεύω και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να εξασφαλίσουμε την επένδυση στους τομείς όπως είναι το, το κυβέρνο έγκλημα και βεβαίως θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο βέλτιστο δυνατό βαθμό στην ανάγκη για συνεργασία, για συμπληρωματικότητα των εργασιών μαζί με τους εταίρους μας και ιδιαίτερα αναφέρομαι εδώ στη συνεργασία με την Όλαφ, με την οποία ήδη έχουμε συζητήσει κάποιες δυνατότητες για συνεργασία. Ιδιαίτερα δε, αναμένω ότι αυτές οι προσπάθειες θα σταθούν με επιτυχία. Αυτό και είναι προσωπική μου δέσμευση τόσο του διευθυντού του Europol όσο και ολόκληρου του προσωπικού της Eurostat. Είμαστε όλοι στρατευμένοι στον αγώνα να καταστεί πιο ασφαλής η Ευρώπη. Και άλλωστε το έχουμε καταγράψει και σε μια προηγούμενη προσπάθεια και συζήτηση που έγινε πρόσφατα. Ιδιαίτερα στοχεύουμε στην καταπολέμηση της ε, διάδοση μέσω του ίντερνετ ε, υλικού σχετικού με κακομεταχείριση παιδιών και ιδιαίτερα σεξουαλική κακομεταχείριση με σκηνές βιασμών ε, ε, και πορνογραφικές σκηνές ε, παιδιών από ηλικία βρεφική κτλ. Έχουμε μαζέψει στο δυνατόν πιο πολύ υλικό και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις μορφές εγκληματικότητας κατά προτεραιότητα. Ευχαριστώ θερμά, λέει η Πρόεδρος. Εγώ σας το λόγο δύο συνάδελφοι. Γεια σας, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Βαρδίνο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα την παρέβασή σας σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 της Europol. Για σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η 23 οι 23 προτεραιότητες που έχετε θέσει αλλά θα ήθελα να θίξω ένα άλλο ζήτημα που ενδεχομένως να γνωρίζετε και αναφέρομαι στο επικείμενο, επικείμενο νομοθετικό έργο που απαιτείται προκειμένου η Europol να ε, ρυθμίζεται μέσω ενός κανονισμού και όχι με απόφαση του Συμβουλίου. Ε, γνωρίζετε και να σας το επαναλάβω ότι το Κοινοβούλιο 17 Ιανουαρίου 2008 ενέκρινε μια τροποποιημένη πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι οι περισσότερες εκ των προτάσεων του Κοινοβουλίου δεν λήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο. Ίσως να μην γνωρίζετε επίσης πως Η απόφαση του Συμβουλίου δίνει κάλυψη νομική στη νέα υπηρεσία του Europol. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010 και στο Κοινοβούλιο δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξει μια νομική κάλυψη μέσω ε, κανονισμού σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα λέω όλα αυτά διότι ο πρώτος στόχος που αναφέρατε έχει σχέση με την ε, ενημέρωση πέραν των ε, όσων ε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και θέλω να σας πω επίσης ότι επήγει το ζήτημα διότι έτσι αναφέρεται και στο πρόγραμμα της Στοχόλμης να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να δουλέψουμε άμεσα για να δοθεί νομική κάλυψη σε μια Europool η οποία θα ε, εντάσσεται και θα υπόκειται στη συνθήκη Λισαβόνα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του προλογούμου κανονισμού στο πρόγραμμα τη και στο πρόγραμμα δράση τη Να σα ενημερώσω επίση πω αύριο πρόκειται να συναντηθώ με τον κύριο Αρμίδα τη Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το θεσμικό ζήτημα. Αυτό μας ενδιαφέρει, διότι το νομοθετικό συγγνώμη ζήτημα. αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τη συνθήκη Αλλά πώ μπορούμε να μιλάμε για κοινοβουλευτικό έλεγχο για αυτό το οποίο εσεί πράτετε σήμερα. Με κάθε σεβασμό που έχω απέναντί σα και απέναντι την παρέμβασή σα. Αλλά αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να ερχόσαστε εδώ να μα εκθέτετε το πρόγραμμα δράση για το 2012 δεν είναι κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι ένας ουσιαστικός κοινοβουλικός έλεγχος που θα στηρίζεται στην ε, Λισαβόνα και στο νέο κανονισμό. Έτσι λοιπόν ε, ε, κύριε Μαρδίνο, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ανάμεσά μας, ευχαριστώ που μας μιλήσατε για το πρόγραμμα εργασιών για το 2012. Ως θα έρθει αργότερα ο κύριος Μπέρν Ράιτ να μας μιλήσει για την εκτέλεση του προγράμματος του 2012. Αλλά αυτό δεν μας πείθει διόλου. Αυτό δεν είναι κοινοβουλικός έλεγχος. Αυτή είναι πληροφόρηση, ενημέρωση. Κάτι το οποίο αξιολογούμε, εκτιμούμε και επιθυμούμε. Αλλά με την βοήθεια της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να θέσουμε σε εφαρμογή τον ε, νέο κανονισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτείνω λοιπόν κύριε Μαρτίνο να ακούσουμε τις ερωτήσεις ε, και μετά να απαντήσετε. Δεν είναι πολλές ούτως ή άλλως, τέσσερις ή πέντε. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Για την, την παρουσίαση για τις δραστηριότητε της Europol. Σας ευχαριστώ επίσης που τονίσατε την σημασία του έργου σας σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, παιδικής πορνογραφίας και κακομεταχείρισης των παιδιών. Αναφερθήκατε επίσης ε, σε ε, θέματα ε, παιδικής πορνείας. Δυστυχώς υπάρχει καταμερισμός εργασιών σε αυτά τα ζητήματα, όπως συμβαίνει και με άλλα αρνητικά φαινόμενα. δηλαδή χρησιμοποιούνται παιδιά από τις νέες, από τις ε, χώρες της Ανατολικής ε, Ευρώπης ε, από κυκλώματα αλλά και όχι μόνο, ακόμα και από στελέχη αν θέλετε, επιχειρημερίες κλπ. Πώς εξετάζετε αυτό το ζήτημα, πώς προσπαθείτε να προλάβετε τέτοιες δραστηριότητες, τι είδους πρόληψη χρησιμοποιείται πολλές φορές. Διαβάζουμε στις εφημερίδες οργανωμένες συμμορίες που συλλαμβάνονται, αλλά δεν ακούμε τη συνέχεια που δίδεται σε αυτό. Έχετε τίποτα success stories να μας πείτε αναφορικά. Άτομα δηλαδή τα οποία φυλακίζονται για μακρό χρονικό διάστημα και τι κάνετε για να προλαμβάνετε τέτοια φαινόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Europol ποιες είναι οι δυσκολίες και τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντάτε προκειμένου να πετύχετε αυτές τις, αυτούς τους κατά στόχους που μας αναφέρατε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, η συμφωνία που υπογράψαμε με τις ΗΠΑ Πολιτείες σχετικά με το TFTP, διότι η Europol είναι ευρωπαϊκή αρχή αρμόδια να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη της συμφωνίας. Δηλαδή από τότε που υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, τι έπραξε η Europol, τι ενημέρωση έχετε σχετικά με την συμφωνία TFTP. Thank you very much, Chair. Um, just briefly, not, not to extend the time, I would just have... Μία ερώτηση. Σε δύο θέματα. που έχουν σχέση με την παράταση της εντολής σας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σύμφωνα με την έκθεση στην οποία αναφερθήκατε, αλλά σε ποιο βαθμό η Ευρωπόλη ήταν ικανή να ασχοληθεί με τα θέματα έγκαιρης προειδοποίησης. Χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλου μεγέθους επιθέσεις οι οποίες δυστυχώς φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν. Έχετε, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων κάποιων ομάδων. Υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με την Ινίσα. Και τι γίνεται, ελπίζω να γίνεται κάτι με το ΝΑΤΟ, γιατί το κέντρο ασφαλείας του ΝΑΤΟ στο Ταλίνα είναι εισμένα λειτουργικό βέβαια, αλλά παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ προσπαθεί να ενισχύσει αυτές τις δομές ασφαλείας του. Λοιπόν υπάρχουν συνέργειες μεταξύ σας. Και δεν ξέρω αν η εντολή σας καλύπτει και το εξής. Κάποια εξτρεμιστικά κινήματα στην Ευρώπη. Είναι τοπικά, εθνικά φαινόμενα Βλέπουμε εξτρεμιστές της δεξιάς της αριστεράς, εγώ δεν κάνω διάκριση εφόσον χρησιμοποιούν βία εις βάρος των αθών. Ή μήπως βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να διασυνδέονται ευρωπαϊκά. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί. Έχετε κάτι για αυτές τις ομάδες, σε πάση περιπτώσει, στα συστήματά σας. τελευταία ερώτηση, δύο τελευταίες τις θέτω εγώ για το κυβέρνο έγκλημα. Όλοι λέγουν ποια είναι τα, ποιες είναι οι απειλές εις βάρος της Ευρώπης. Αλλά οι ισχυρισμοί αυτοί βασίζονται σε εκθέσεις εταιριών όπως η Symantec που έχουν ζωτικά ε, επιχειρηματικά συμφέροντα. Γνωρίζουν πολλά πράγματα αλλά παρόλα αυτά έχουν συμφέρον εδώ γιατί πολλούν συστήματα ασφαλείας σας λένε ότι υπάρχουν απειλές και σας πουλάνε τα συστήματα ασφαλείας σας. Δεν αμφισβητώ εγώ την ποιότητα των εκθέσεων, αλλά μήπως θα χρειαζόμασταν κάποιες πιο ανεξάρτητες αξιολογήσεις της κατάστασης. Δεύτερη ερώτηση, πάντα για το κυβερνοέγκλημα. Προσπαθούμε να δούμε τι θα έκαναν οι εγκληματίες του διαδικτύου εις βάρος των κυβερνητικών ηλεκτρονικών δομών κτλ αλλά και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες είμαστε πάρα πολύ θα έλεγα ευάλωτοι και πολλές φορές τα συστήματα προστασίας που έχουμε δεν τα καταφέρνουν. Σαν παράδειγμα το κίνημα ανώνυμους ε, την προηγούμενη εβδομάδα δημιούργησε πολλά προβλήματα και έριξε τα συστήματα του FBI και της CIA. Εσείς ελέγχετε τα δικά σας συστήματα, επειδή συλλέγουμε συνεχώς όλο και περισσότερες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, είναι προστατευμένα τα δεδομένα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Lisbon Treaty. Καθώς ερχόμουν εδώ, αναρωτιόμουν ποιος είναι ο λόγος, είναι σωστότερος έλεγχος, είναι οι πληροφορίες. Εσείς βέβαια είστε το σώμα το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό μας και εφόσον εγκρίνετε τον προϋπολογισμό μας έχετε κάποιο έλεγχο ε, σε μας. Ταυτόχρονα θα μπορούσατε να μας προσκαλέσετε να σας δώσουμε και τα επιχειρηματικά μας σχέδια, τους στόχους μας, τις προτεραιότητές μας. Και ιδιαίτερα τον προγραμματισμό μας για το 2013, ο οποίος μόλις ενεκρίθη από τη Διαχειριστική Επιτροπή και περιμένουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα υιοθετηθεί το φθινόπωρο του 12, ίσως πριν να ζητήσετε από τον εκπρόσωπο του Ευρωπόλ της Ευρωπόλ να σας πει τι σκοπεύουμε να κάνουμε του χρόνου. Εσείς λοιπόν θα θέσετε ερωτήσεις, πρέπει να θέσετε ερωτήσεις. Εγώ σήμερα σας δίνω κάποιες πληροφορίες ε, για το τι συμβαίνει φέτος που βρισκόμαστε στο τέλος του δεύτερου μήνα. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς απέναντί σας, θέλουμε να μοιραστούμε τις προτεραιότητές μας θέλουμε να συνταυτιστούν θα έλεγα μέσω του προϋπολογισμού που παίρνουμε οι πολιτικές μας, να βασιστούμε στον κύκλο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί τη βάση των αποφάσεων βέβαια που λαμβάνει τα, οι το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ευρωπόλη είναι υπεύθυνη για θέματα εφαρμογής, θυμίζω. Εμείς δεν δημιουργούμε πολιτική, δεν γεννάμε πολιτική. Βέβαια φυσικά λέμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας για κάποιες βελτιώσεις των δραστηριοτήτων μας κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες, δεν είμαστε ιδιοκτήτες των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες ανήκουν στα κράτη-μέλη και μπορούμε να πάρουμε μέρος στις διαδικασίες αυτές. Και οι απόψει σας, ιδιαίτερα οι δικές σας απόψεις σαν κοινοβουλευτικό σώμα είναι καλοδεχούμενες. Αυτά τα λέω για την ερώτησή σας τη σχετική με το νέο νομικό πλαίσιο. Και σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης τώρα, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, η εφαρμογή αυτού του νέου νομικού πλαισίου θα πρέπει να αξιολογηθεί. Η εταιρεία Rent Europe έχει επιλογή. Έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες εκθέσεις. Την Ιούνιο περιμένουμε την τελική έκθεση η οποία θα μας βοηθήσει να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση για την Ευρωπόλ στο μέλλον. Προσπαθούμε να προσθέσουμε αξία θα έλεγα στις ερευνητικές διαδικασίες ε, τις οποίες διεξάγουν τα κράτη-μέλη. Τέθηκε επίσης το θέμα της TFTP. Uh, Η συμφωνία λοιπόν τη FTP. Καλή ερώτηση αυτή. Προφανώς συνεργαζόμαστε στενά με το σώμα αυτό, το ελεγκτικό, το οποίο συνεδριάζει συχνά και ο ρόλος της Ευρωπόλ είναι και να ελέγχει ελέγχοντας ότι τα αιτήματα των Αμερικανών είναι συμβατά με το περιεχόμενο της συμφωνίας που έχουμε μαζί τους. Αν θυμάμαι καλά, λάβαμε 14 αιτήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η Europol έλεγξε τα αιτήματα αυτά και τα ενέκρινε. Send several requests to και ταυτόχρονα στείλαμε αρκετές, αρκετά αιτήματα από τις Ηνωμένε Πολιτείες και πήραμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικές με τις ερευνητικές δραστηριότητες των κρατών μέλων. Δεν μπορώ να σας δώσω ε, περισσότερες πληροφορίες γιατί οι πληροφορίες αυτές αφορούν ε, έρευνες οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή σχετικά με ομοκρατικές επιθέσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Πάντως ο ρόλος της Ευρωπόλ είναι να ελέγχει τα αιτήματα αυτά. Δεν έχουμε εμείς πρόσβαση στις ίδιες τις πληροφορίες οι οποίες αποστέλλονται στις Ηνωμένε Πολιτείε μέσω του SWIFT. Αυτά σχετικά με το TFTP. Και τώρα, η Κοινή Ελεγκτική Επιτροπή δημοσιεύσε την, ε- δημοσιεύσε την έκθεσή της ή μάλλον θα δημοσιεύσει την έκθεσή της στο τέλος Μαρτίου για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Πολύ καλή ερώτηση. Θα συμφωνώ όμως με την Πρόεδρε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι, ιδιαίτερα σαν χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πηγαίνουμε και ελέγχουμε κάτι στους υπολογιστές μας και μερικές φορές βλέπουμε ότι ο υπολογιστής μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στρεβλά από αυτούς που είναι επιφορτισμένοι να μεταφέρουν σαν παράδειγμα πληροφορίες ε, σε σχέση με δραστηριότητες όπως το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος. Οι υπολογιστές μπορεί να χρησιμοποιηθούν με κακούς στόχους, να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να ευαισθητοποιήσουμε τους χρήστες. Και φυσικά εδώ οι κατασταλτικές μονάδες, δυνάμεις μάλλον, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες, να συλλέγουν στοιχεία, να μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά στα δικαστήρια, να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν αν θέλετε αυτούς οι οποίοι παρανομούν. Αυτή είναι η υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε. Εμείς μπορούμε να παίξουμε ηγετικό ρόλο, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τον έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ποια είναι η ανώτατη αρχή αν θέλετε. Πάντως η Ευρωπόλ μπορεί και θέλει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο όπως είπα. Η δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με την ίδια την Ευρωπόλ και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει. Η θέση μου είναι συντονιστής ασφαλείας στην Ευρωπόλ και μετά από τις επιθέσεις των ανώνυμους ξεκινήσαμε ένα εκ νέου έλεγχο των ρυθμίσεων ασφαλείας μας στο εσωτερικό της Europol, πώς οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε κρατούνται σε εισαγωγικά με ασφαλή τρόπο και θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια. Ζούμε στον κυβερνοχώρο, δεν μπορούμε να μείνουμε εκτός κυβερνοχώρου. Είμαστε υπεύθυνοι για την καταπολέμηση φυσικά σε πολλούς τομείς του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και είμαστε υπεύθυνοι και για να ελέγχουμε εσωτερικά τις δικές μας δυνατότητες και τις δικές μας άμυνες. Πάντως μέχρι τώρα χτυπάω ξύλο. Τα πράγματα πάνε καλά, δεν, είχαμε, δεν έχουμε υποστεί επιθέσεις ιδιαίτερες και τα δεδομένα που έχουμε στις, ε, στις τράπεζες δεδομένων που διαχειριζόμαστε είναι ασφαλή πάντα. Δεν έδωσα απαντήσεις νομίζω σε όλες τις ερωτήσεις. Το αίτημα για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τα επιπλέον βήματα που πρέπει να κάνουμε Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς ακριβώς ε, ε, προχωρούν οι διαδικασίες σχετικά με το ποινικό δίκαιο. Απαιτείται κάποιος χρόνος, δεν είναι θέμα εβδομάδων απλά. Μερικές φορές χρειάζεται πάνω από ένα χρόνο για να μπορέσουν κάποιες περιπτώσεις. Προφανώς αναφέρεται σε θέματα βιοπαγιών εις βάρος παιδιών. Ο μιλητής. Ε, για επιμέρους θέματα στα οποία ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες για το πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες, οι ανακρίσεις, οι έρευνες και τι αποτελέσματα έχουμε στο τέλος. Καλώς ευχαριστώ, λέει η κυρία Ιντβελτ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και βεβαίως θα ακούσουμε και την υπόδειξή σας. Όπως και εσείς. Του κύριου Διασδεμίρα για πιο ουσιαστική δημοκρατική επιτήρηση. κυρία Χάνκης από ό,τι μαθαίνω τώρα δέχεται το θέμα της, που είναι το τελευταίο της σημερινής ημερησίας διάταξης, να το συστήσουμε αύριο το πρωί, κάπου στις 11. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε στα σημεία 5 και 6 της σημερινής διάταξης, με παρουσία της κυρίας Λεμπάη. Σημεία 5 και 6 λοιπόν, προστασία των ιδιωτών σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διακίνηση προσωπικών δεδομένων, δηλαδή κανονισμός, γενικός κανονισμός για προσωπικών δεδομένων και στο σημείο 6 προστασία των ιδιωτών σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές με στόχο την πρόληψη, διαρεύνηση, άνοιχνευση ή δίωξη Ε, εγκληματικών ε, δραστηριοτήτων ή την, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Θα ακούσουμε όμως πρώτα την κυρία Λεμπάγε, Γενική Διευθύντρια για θέματα δικαιοσύνης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Επιτρέψαμε να προβάσω μια γενική παρουσίαση των δύο μέσων μαζί των δύο νομοθετημάτων, γιατί ε, πιστεύω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική υπό την οποία επιλέγει την παρού, ταυτόχρονη παρουσίαση των δύο αυτών νομοθετημάτων. Και επιτρέψτε μου καταρχάς να υπογραμμίσω το πλαίσιο στο οποίο καταθέτουμε αυτές τις προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, η νομοθεσία μας οδηγεί ακόμα έχει ηλικία 17 ετών, με ένα μόνο τη 100 την εποχή εκείνη της χρήση ε, του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον ε, πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε πόσο ριζικά έχει αλλάξει η κατάσταση ε, έκτοτε και πόσο απαραίτητη καθίσταται μια ανανέωση, μια αναθεώρηση της νομοθεσία. Επίσης, η φύση του, νομοθετήματο, νομοθετήματος, η οδηγία, ως εκφύσεω έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύ κατακαιρματισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 διαφορετικά καθεστώτα προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει από τα κράτη-μέλη και άρα πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση ακριβώς λόγω του κατακαιρματισμένου ε, της εφαρμογής και της ανάπτυξης μέσων τα οποία μπορεί να ήταν χρήσιμα πριν από 17 χρόνια αλλά που 17 χρόνια αργότερα καλούμε, θα βλέπουμε απαραίτητο να αναθεωρήσουμε. Αλλά πάντω κέριο ο ρόλο, στην υπόθεση αυτή να όλοι έπεσε, έπαιξε και η συνθήκη τη Λισαβόνα, η, οποία, η οποία υπό το άρθρο 16 ε, ορίζει ρητά ότι ο καθένα έχει δικαίωμα στην προστασία του προσωπικού του δεδομένων, άρα μετατρέπει, αναγνωρίζει τα, τα προσωπικά δεδομένα ω σε δικαίωμα και άρα είμαστε υποχρεωμένοι να ε, υποταχθούμε και εμείς αυτήν την επιταγή και την προοπτική. Η οδηγία λοιπόν αντίστοιχες με την πρώτη οδηγία είχε και η οδηγία σχετική με τον δικαστικό τομέα, απόφαση πλαίσιο, που είχε σε ένα αποτέλεσμα πολύ διαφορετική εφαρμογή αυτής της οδηγίας της απόφασης πλαισίου από το ένα κράτος μάλλον στο άλλο. Και έτσι με δεδομένα όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταθέσει μια πρόταση με τη μορφή δέσμης, με ανακοίνωση καταρχάς, δεν σας κατέπληξε ασφαλώς, διότι είχαμε προεξαγγείλει ένα χρόνο πριν στην ανακοίνωσή μας για την που των θα παίρνουν την πρόθεση αυτή. Αλλά ανακοίνωση και δύο νομοθετήματα πρώτα απ' όλα με αλλαγή ως προς τον κανονισμό στη μία περίπτωση και δεύτερον ως προς την οδηγία στην άλλη. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να σας εξηγήσω τι προσπαθούμε να πράξουμε. Τι επιτυχάνουμε, προσπαθούμε να επιτύχουμε με την ε, υποβολή αυτών των προτάσεων. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ιδιωτών και αυτό εύλογα, διότι μετά από μια διαδικασία διαβουλεύσεων στην οποία είχαμε και ε, επί διετία ε, διαβουλεύσεις με εμπλοκόμενους φορείς κάθε είδους, διαπιστώσαμε ότι είδαμε και τις απόψεις του Κοινοβουλίου με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θελήσαμε ασφαλώς να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ιδιωτών. Η ενίσχυση λοιπόν των δικαιωμάτων των ιδιωτών πρέπει να περάσει από έναν τρόπο, από μια μεθοδολογία η οποία θα εξασφαλίζει στον ιδιώτη δικαίωμα να μένει στα αζήτητα τρόπον την. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει κανείς να έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα προσωπικά του δεδομένα. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και να μην τον θυμάται κανείς, να μένει στα αζήτητα. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει καμία επέμβαση ή περιστολή του δικαιώματος στην, ε, λόγο, στην ελευθερία της έκφρασης. Απλώς προσπαθούμε το δικαίωμα του να μένει κανείς στα αζήτητα και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης να αξισορροπηθούν και να σταθμιστούν σωστά. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, προσδορίσουμε και την έννοια της συνένεσης όταν ζητείτε, απαιτείται συνένεση όταν στείτε μάλλον η συνένεση από τον ιδιότητα, πρέπει, ε, από τον ιδιότητα αυτός πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνει αυτή η συνένεση και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί ε, θα συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να αντιληφθεί κανείς τι ε, συνέπειες μπορεί να έχει η συνένεση που του ζητείτε. Δικαίωμα στην πληροφόρηση επίσης, δηλαδή πρέπει να γνωρίζει κανείς τι τύχη θα έχουν τα δεδομένα του εφόσον δώσει τη συνένεσή του και εφόσον αυτά στη συνέχεια περάσουν από μια ε, επεξεργασία από οργάνωση ενδεχομένως ιδιωτική εταιρεία αφενός, αλλά και δημόσιο φορέα αφετέρου πιθανώς. Θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα του ιδιώτη. Αλλά ταυτόχρονα η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει εξυπαρχής. Όταν δηλαδή μια επιχείρηση, μια εταιρεία αναλογίζεται την εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας, ήδη να λαμβάνεται υπόψη. Και γι' αυτό μέσα στον κανονισμό θα αναγνωρίσετε φαντάζομαι την έννοια της προστασίας των δεδομένων εκ των προτέρων, ε, που σημαίνει ότι όταν σχεδιάζει κανείς μια νέα διαδικασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να προβλέπει τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πράγμα, είναι το πολύ, πράγμα το οποίο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και οικονομικό από το να προσπαθήσει κανείς εκ των υστέρων να αντιμετωπίσει παραβιάσεις ενδεχομένω των προσωπικών δεδομένων. Και ζητούμε από τις επιχειρήσεις να ορίζουν ε, σε μεγάλες επιχειρήσεις βέβαια ε, άνω των 250 εργαζομένων κάποιον, ε, κάποιος τέλεχος αρμόδιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εισάγουμε και την έννοια της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, άρα βλέπετε σημαντική ενίσχυση των δικαιωμάτων των ιδιωτών. Ένα άλλο πολύ ξεκάθαρο στοιχείο πιστεύω που θα στην ε, πρόταση κανονισμού είναι η πολύ σαφής παρουσία της ενιαίας αγοράς. Όπως είπα, με φόντο τα 27 διαφορετικά καθεστώτα, προσπαθούμε να εισαγάγουμε μια ενιαία νομοθεσία, μια ε, ενιαία τοποθέτηση. Άρα δηλαδή ενιαία νομοθεσία γιατί ο κανονισμός εξορισμού δεν χρειάζεται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, έχει άμεση εφαρμογή και ως εκ τούτου μόνο ένα νομοθέτημα θα ισχύει για τον κάθε ένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, με τεράστια πλεονεκτήματα και ωφέλη στην οικονομία μας, γιατί συνεπάγεται εξοικονόμηση 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ή ύπαρξη ενός μόνο καθεστώτος νομοθετικού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προπητήρουμε επίσης μια μονοθυριδική προσέγγιση. Μια επιχείρηση δηλαδή θα έχει μόνο μία αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την οποία θα έχει να συνδιαλλαγεί. Ε, πράγμα το οποίο αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα, ότι δεν ήξερε κανεί με ποια αρχή προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να συνδιαλέγει, αν θα έπρεπε να απευθυνθεί στην εθνική του αρχή προσωπικών δεδομένων ή την αρχή προστασία των προσωπικών δεδομένων στο κράτο μέλο του οποίου, στο οποίο, στο οποίο έχει την έδρα της η επιχείρηση. Και γι' αυτό λοιπόν, για να το αποφύγουμε αυτό, θεσπίσουμε μια μονοθυριδική προσέγγιση με την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων στο κάθε κράτο μέλο ω αντιπιστέλων μέλο. Και έτσι έχουμε και το δικαίωμα για τον ιδιώτη που ταυτόχρονα ενισχύει την απλούστευση, την απλοποίηση στην ενία αγορά. Ας ε, αναφερθώ λίγο σε αυτό. Είχαμε δεκάδες χιλιάδες προσπάθειες απλοποίησης στον τομέα της ε, ε, προστασίας των δεδομένων και μόνο σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις δεχόμαστε τις διαδικασίες, αλλά έχουμε εισαγάγει μαζικές απλοποιήσεις στον τομέα των προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά λοιπόν απλουστεύουν και ταυτόχρονα ενισχύουν, απλουστεύουν το σύστημα, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν και την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Και ξέρετε ότι πολλοί είναι οι καταναλωτές εκείνοι οι οποίοι αποφεύγουν να ψωνίσουν, να μπουν δηλαδή σε μια ιστοσελίδα για να αγοράσουν προϊόντα υπηρεσίε, γιατί πρώτα δεν γνωρίζουν τι μοίρα μπορεί να έχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και πώς θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Και επίσης δεν γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν σε περίπτωση διάρρηξης του συστήματος ε, της επιχείρησης του φορέα που έχει αναλάβει την ε, ε, διαχείριση των δεδομένων αυτών. Και εδώ προτείνουμε μια σαφέστερη και πιο αυστηρή διαδικασία κοινοποίησης με 24 ώρες βάσης δυνατότητα υποδοχής ε, ενημέρωσης, κοινοποίησης για τέτοιες ε, παραβιάσεις και βέβαια με ένα σαφή κατάλογο τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να ενημερωθεί ο εμπλεκόμενος ιδιώτης, εκείνος δηλαδή του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν παραβιαστεί ε, ε, εν ευθέτω χρόνο. Μονοθυριδική προσέγγιση, μία νομοθεσία, απλούστευση, όλα αυτά φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά όμως πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη. Πιστεύω ότι και πάλι με μία θαραλέα προσέγγιση αναπτύσσουμε έναν μηχανισμό συνέπειας, καταρχάς για να μην επιμένω σε αυτό, προσπαθούμε, ε, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις αρχές προστασίας των δεδομένων, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ε, ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει κάθε αρχή προστασίας των δεδομένων και αυτό περιμένουμε να δούμε να συμβαίνει. Και εν προκειμένου θέλουμε ε, προστασίες δεδομένων με κοφτερά δόντια, δηλαδή να έχετε δυνατότητα η κάθε υπηρεσία προστασία δεδομένων να επιβάλλει πρόστιμα υψηλά, πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης, τα οποία θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Ναι, έχω ακόμα τρία λεπτά, ευχαριστώ. Ε, για την προστασία λοιπόν των δεδομένων φαντάζεστε ότι μπορώ να μιλάω ε, ασταμάτητα. Λοιπόν, θα περιοριστώ όμω τα τρία λεπτά. Ενισχύουμε λοιπόν τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Έχουμε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τις διαφορετικές ερμηνείες του νόμου που ενδεχομένως να προκύπτουν όταν εμφανίζονται νέα τεχνολογικά μέσα. Φερρυπίν, στο Google Street View αυτό που συνέβη. Και έτσι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια ε, ως το δυνατόν ενιαία ε, ερμηνεία των ε, διατάξεων της νομοθεσίας. Και το τελευταίο κομμάτι που αφορά τον κανονισμό έχει να κάνει με τις διεθνείς μεταφορές στοιχείων. Τι συμβαίνει εκεί. Προσπαθούμε να προσθέσουμε την κατάσταση. Όταν έχουμε μέσα σε ένα μεγάλο όμιλο εταιρικό μεταφορά δεδομένων. Προσπαθούμε να ε, την παρακολουθήσουμε, προσπαθούμε να έχουμε σαφείς κανόνες καταλληλότητα στη μεταφορά και γενικά κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτά για τον κανονισμό. Και πολύ σύντομα, δεν θέλω να πω δύο λόγια για την οδηγία σχετική με την αστυνομία. γιατί να προτείνουμε οδηγία. Ενώ έχουμε πρόταση κανονισμού για τα εμπορικά δεδομένα. Να σα πω δύο ότι ο τομέα τη αστυνομία και τη δικαστική συνεργασία είναι ένα ευαίσθητο τομέα και βεβαίω απαιτείται να έχουμε και θέλουμε να έχουμε προσθέτει ευελιξία στο τομέα αυτό. Σημαντικό πάντως είναι το ότι έχουμε εξασφαλίσει ένα σημαντικό βήμα προόδου. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε σε κάθε βήμα ε, την οδηγία και δεύτερον γιατί θέλουμε να έχουμε μια διαδικασία ε, στο εσωτερικό που δεν προβλέπεται από την οδηγία. Και όταν υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, εξαιρέσεις από τον τομέα αυτόν, πρέπει τα κριτήρια για τις εξαρτήσεις αυτές να είναι εναρμονισμένα μεταξύ των κρατών μελών. Mm. Αυτά με αδρές γραμμές και παραλαμβάνω θα μπορούσα να μιλάω ώρες ακόμα. Είναι μια θαραλέα μεταρρύθμιση, αυτή που σας παρουσιάζω, μια μεταρρύθμιση η οποία εξασφαλίζει πολύ περισσότερα πράγματα για τα δικαιώματα των ιδιωτών από ό,τι έχουμε τώρα για μια μεταρρύθμιση η οποία προστεύει επίσης σημαντικά και ενισχύει την εσωτερική αγορά, εξασφαλίζοντας εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, που έχει κέρια σημασία για την ανάπτυξή μας, ενώ ταυτόχρονα προτείνουμε την απλούστευση για τις διεθνείς μεταφορές στοιχείων. Αυτά ε, έχουμε ξεκινήσει την συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου με πρώτη συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα και αναμένουμε τη συνέχιση των εργασιών και την ανάληψη συνομιλιών με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Με έκπληξη είδα ότι την προηγούμενη ομάδα οι Αμερικανοί εταίροι μας απέστειλαν μήνυμα ότι και εκείνοι θεωρούν πως ε, είναι σωστή επιλογή μιας, ε, μια ολιστική επιλογή για την προσέγγιση, μια γενική δηλαδή προσέγγιση, ενώ μέχρι τώρα είχαν διαφορετική αντίληψη, αλλά φαίνεται ότι έχουν ε, αλλάξει στάση, πάνε προς το σωστό δρόμο που είναι βεβαίω ευρωπαϊκός. Και πάλι πιστεύω μπορούμε να εξασφαλίσουμε χάρη σε αυτή την ε, αλλαγή και των Αμερικανών μια καλή αποτελεσματική προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολύ ώρα. Πράγματι είναι πολύ κομβικό το θέμα. Five requests for the floor, including myself. Are there any six? Okay, okay. You take the names. Um, I suggest we take them uh, three by three. Uh... Ανά τρεις ερωτήσεις ε, θα την χάνουν απαντήσεων από πλευρά σας. Παρακαλώ συνάδελφοι όμως να μην ξεπερνάτε το χρόνο σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ την κυρία Λεμπάη. Πράγματι, έχει γίνει τεράστια προσπάθεια, δεν ήταν εύκολο να δημιουργήσει κάτι το οποίο χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο για να υπάρξει. Παρ' όλα αυτά έχουμε φτάσει τώρα πια στη διαδικασία αναθεώρησης της πρότασης και όπως είπατε υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συναδέλφων που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή γιατί δεν υπερβάλλω, αυτός ο κανονισμός ίσως είναι από τους πιο σημαντικούς σε αυτή την περίοδο. Είναι ένας από τους λίγους κανονισμούς που επηρεάζει όλο τον κόσμο και αυτούς που είναι εδώ και αυτούς που είναι εκτός και στο Βέλγιο και εκτός Βελγίου, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Γι' αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε κάτι στη διάθεσή μας το οποίο να καλύπτει αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα κριτήρια τα οποία να συμφωνούν με τη λογική της πρότασης, ε, με... να δούμε πρακτικά τι υπάρχει, τι λείπει υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν. Σαν παράδειγμα, στις αιτιολογικές σκέψεις ακούγονται πολλά για τη διαφάνεια, τα οποία όμως δεν φαίνονται στα άρθρα και αυτά δημιουργούν μια μικρή σύγχυση στην εφαρμογή όπως είδαμε ε, και σε άλλες αντίστοιχες οδηγίες. Περαιτέρω, στις αιτιολογικές σκέψεις ε, ο καθορισμός των προσωπικών δεδομένων αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια φαιά περιοχή. Το θέμα είναι όμως ότι σε επίπεδο άρθρων δεν διευκρινίζεται απόλυτα νομικά η κατάσταση και εκεί δημιουργείται μια επιπλέον σύγχυση. Ε, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ο κανονισμός αυτός δεν είναι ένας κανονισμός Facebook ή κανονισμός Google, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να καλύψει αν θέλετε ε, όλους οι οποίοι ασχολούνται με θέματα αυτά, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι ε, δικηγόροι. Ξέρουμε ότι το 95% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών έχουν πολύ λιγότερους από 200 εργαζομένους για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ξέρετε ότι και εδώ ε, πρέπει να κάνετε μία πρόταση η οποία δεν θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει κατά 80% μέσω ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μένει να γίνουν. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και μαζί σας και με την Προεδρία γύρω από το θέμα αυτό. Ο Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και τις καλές εξηγήσει. Γνωρίζουμε ότι η οδηγία του 95 είναι καλή και έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και να επικρινώ ο κανονισμός και η οδηγία. Νομίζω ε, αντικατοπτρίζουν σωστά την, ε, κατανομή των τομέων ε, και άρα θα έλεγα ότι επί τη βάση των όσων έχουμε να συζητήσουμε, θα έλεγα ότι πολύ ικανοποιημένοι συνόμαστε για το πρώτον σε πόσο βαθμό έχουμε προχωρήσει, την πρόοδο που έχει σημειωθεί, και δεύτερον αυτά που σκοπεύετε να κάνετε. Η έκθεση πρωτοβουλία που είχαμε το φθινόπωρο άλλωστε είχε υπογραμμίσει και τα ίδια, δηλαδή πλήρη εναρμόνιση, ασφάλεια δικαίου για πολίτε ε, και επιχειρήσεις, ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και εκτός του δημοσίου χώρου, δυνατότητα διόρθωση ε, απάλληψη κτλ. Όχι μόνο πρόσβαση. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν τα οποία είχαμε ζητήσει έχουν γίνει δεκτά και ευχαριστούμε θερμά. Από την άλλη, κάποια σημεία ασφαλώ θα χρειαστούν περαιτέρω συζήτηση, διόρθωση, προσαρμογή, διευκρίνηση. Ίσως χρειάζεται να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Και πάντως πρωτεβλέπουμε ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να μην θα πρέπει πάντοτε να προχωρούν με σεβασμό των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου και των προνομιών, όπως είπε και ο κύριος Άλβαρο. Θα πρέπει να δούμε στην περίπτωση των, των κοινοποιήσεων σε κάποια περίπτωση παράβασης ε, πώς λειτουργεί το σύστημα και ε, κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση και με το cloud computing. Αυτά δεδομένου δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα απλώ να επισημάνω ότι θα μα απασχολήσει το θέμα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Άλμπρεχτ, αλλά πολύ σύντομα μου επιτρέπετε, ε, δέχεστε να ακούσουμε όλε τι ερωτήσει, μια και είναι μάλλον γενικού χαρακτήρα και όχι τεχνικού, και μετά να απαντήσετε. Ο κύριο Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, την κυρία Λεμπάγιο. Πιστεύω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τα μέχρι τώρα σχόλια. Ήταν καλή αυτή η πρώτη πρόταση που είδαμε, μας ε, προσφέρει μια καλή βάση εργασίας και σημαντικό είναι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά βέβαια και στο Συμβούλιο των Υπουργών από κοινού να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για την τελική μορφή που θα λάβει ο κανονισμός. Πιστεύω δε επίσης ότι υπάρχουν και κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει πιο διεξοδικά να συζητήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως υπόθηκε άλλωστε είναι ο τομέας των ουσιαστικών αποφάσεων που θα θέλουμε να λάβουμε σε σχέση με τον κανονισμό. Βεβαίω είναι ένα αρκετά ριζικό νομοθετικό μέσο ο κανονισμός και γι' αυτό θα, πρέπει να ορίζεται ξεκάθαρα το τι ρυθμίζει για να εξασφαλίζει και την ασφάλεια δικαίου και άρρωση εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ορισμοί, πολύ πιο σαφείς ορισμοί και στην περίπτωση των κατεξουσιοδότησης συμπράξεων που προβλέπονται πάλι θα πρέπει να κάνουμε την διαφοροποίηση όταν είναι κάπως σαφής η διατύπωση ε, ή όταν μπορεί ο νομοθέτης να δώσει πολύ πιο συγκεκριμένους όρους εφαρμογής ή όπου μπορεί να δώσει ενδεχομένω κάποιο πεδίο ε, το οποίο θα ανήκε ακόμη στο πεδίο ρύθμιση των κρατών μελών, νομοθετική παρέμβαση των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι μπορούμε από κοινού να εξασφαλίσουμε ένα σαφέστερο και πιο ισχυρό πεδίο προστασία των προσωπικών δεδομένων των ε, ιδιωτών, όπω απαιτεί το Κοινοβούλιο παγίως mm. και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάθε ένα σημείο αυτής της ε, προτάσεως να τα συζητήσουμε ένα-ένα, να δούμε τι χρειάζεται τροποποίηση, να δούμε τι μπορεί να μείνει όπως έχει και βεβαίως περιμένω πολύ καλή συνεργασία και με τους ε, της ε, Συμβούλου και Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις βασικές διατάξεις που είναι το δικαίωμα του να ξεχαστεί και το ζήτημα της ε, συνένεσης. Είχαμε, ξεκινήσαμε κάποιες συζητήσεις ε, με τους υπεύθυνου και θέλω να γνωρίζω κατά πόσον έχουμε πετύχει μια κατάλληλη ισορροπία εδώ, μη σωστή ισορροπία για το θέμα της ψηφιακής οικονομίας που θέλει να είναι μια πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Έχα διάφορες εταιρείε telemarketing και άλλες με τις οποίες συνομίλησα και που ανησυχούσαν ότι θα δημιουργήσουμε ε, περισσότερη γραφειοκρατία. Αλλά παράλληλα θέλουμε και οι ιστοσελίδες να λειτουργούν ε, αποτελεσματικά, να υπάρχει δυνατότητα επιγραμμικών αγορών ε, και οι μεταφορές που έγιναν μετά από συνένεση και Τι γίνεται όταν ε, προσπαθούν οι επιχειρήσεις ε, να βρουν ή να αναζητήσουν δεδομένα. Θα υπάρχουν κατευθυντές γραμμές. Ε, πώς θα λειτουργούσουν. Υπάρχει και το ζήτημα των DPA στις χώρες. Πώς θα λειτουργήσουν λοιπόν όλα αυτά στην πράξη. Η Κομισιόν σίγουρα τα έχει σκεφτεί όλα αυτά. Ξέρω ότι θα ασκηθούν πολλές πιέσεις ε, και θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν καταστάσεις ενδιαφερόμενων, ε, και φυσικά υπάρχουν και τα cookies ε, τα οποία υπάρχουν στην θεωρία αλλά και στην πράξη. Ευχαριστώ κυρία Βέρζα. Κυρία Βέρζα, παρακαλώ, έχετε λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, είπατε κύριε Γενική Διευθύντρια, το ψηφιακό περιβάλλον έχει εξελιχθεί σημαντικά τελευταία, πρέπει να προσαρμοστεί. Γι' αυτό λοιπόν θα αναφέρω κάποια στοιχεία. Γιατί δύο κείμενα. Μας είπατε, αλλά η εξήγησή σας ε, δεν με ικανοποίησε. Ειδικά όταν λέτε πως χρειαζόμαστε ευελιξία. Η οδηγία σημαίνει δυνατότητα προσαρμογής για τα κράτη-μέλη και γνωρίζουμε πως ε, αυτό το ζήτημα η νομοθεσία σε δικαστικά ζητήματα χρησιμοποιείται μαζικά από τον πληθυσμό με τρόπο δυσανάλογο σε σχέση με τον στόχο. Εάν λοιπόν υπάρχει οδηγία τότε τι εγγύησεις θα έχουμε για αυτού του είδους την διολίστηση όταν γνωρίζουμε ότι σε ό,τι φορά την παραβίαση των θεμελιών δικαιωμάτων τα κράτη-μέλη κρύβονται πίσω από την αρχή της επικουρικότητας. Το θλιβερό παράδειγμα της Ουγγαρίας μας το αποδεικνύει περίτρανα. Ποιο θα είναι ο λόγος του Ευρωπαίου επόπτη προστασία δεδομένων γιατί τι διάρθρωση θα έχει με τον νέο οργανισμό που πρόκειται να συστηθεί, που θα αντικαταστήσει την Επιτροπή Άρθρου 29, που όντως ε, ζητούσε να αποκτήσει ένα καθεστώς κατάλληλο του ονόματος. Ε, κάτι ακόμα. Έχουμε ανησυχίες σχετικά με το άχθος των επιχειρήσεων. Δεν θα υπάρχουν πλέον ε, εκ των προτέρων διαδηλώσεις παρά μόνο αν ε, προκύψουν σοβαρές παραβάσεις. Και δεν με ικανοποιεί τίποτα από όλα αυτά, διότι όλοι νομίζω ότι στηρίζονται στην καλή ενημέρωση των πολιτών και διαρωτώ με ε, το, τι γίνεται με το ζήτημα των πλέον ευάλωτων πολιτών, τι προστασία θα έχουν. Και δύο ακόμα ερωτήματα Κυρία Βερζά, κύριε Βερζά, δύο λεπτά είχα τη διεύθυνση σας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, γρήγορα, Πρόεδρε. Το άρθρο 29 της οδηγίας αναφέρει πως ε, οι προηγούμενες οδηγίες θα παραμείνουν αμετάβλητες. Ε, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά το πώς θα γίνουν όλα αυτά και το άρθρο 69 για τις ε, αιτήσει διεθνούς τροποποίησης, πώς ε, ρυθμίζουμε το ζήτημα PNR, PNR των είπαν όταν αναφέρουμε, αναφέρεται πως ε, τα, κάποια διεθνή άρθρα πρέπει να τροποποιηθούν. Κυρία Ρομέρο Λόπεζ, ευχαριστώ. Να τονίσω πως ο κόσμος όντως άλλαξε, οι ε, διαφοροποίησαν τον κόσμο μας, ε, αλλά οι νέες τεχνολογίες ε, μας οδηγούν σε μια δίωξη δικαστική, αστυνομική θα έλεγα. Και το είδαμε αυτό στην συμφωνία που συζητήσαμε προ λίγο και θα ψηφίσουμε για το PNR. Θα δούμε λοιπόν εάν ε, το άρθρο της οδηγίας υπαρθμών 9 και το άρθρο 10 παραβιάζουν η αδίποτε κατάχρηση κατά την επεξεργασία δεδομένων και την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν κάποιες προσωπικές ε, πτυχές, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ γενικόλογο ως διατύπωση. Αυτές οι συμφωνίες που υπογράφουμε παραβιάζουν αυτή την οδηγία προστασίας δεδομένων. Διότι τότε εδώ κάνουμε τα πράγματα στραβά. Υπογράφουμε μια συμφωνία για PNR και τώρα φτιάχνουμε την οδηγία για προστασία δεδομένων. Ανάποδα πάμε. Βάζουμε πρώτα τη σκεπή και μετά τα θεμέλια. Το άρθρο 2 λέει ποιος είναι ο στόχος που βρίσκεται εκτός, εκτός οδηγίας. Είναι η εθνική ε, ασφάλεια. Αλλά το πεδίο εφαρμογή αυτών των διεθνών συμφωνιών δεν αφορούν την, ε, την ε, εθνική ασφάλεια, είναι τρομοκρατία, οργανωμένο, σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, διασυνοριακό κλπ. Τι θα γίνει λοιπόν, θα, παρα, θα παραβιάσουμε την οδηγία αυτή. Αυτή είναι μια αφιβολία που με ταλανίζει αυτή τη στιγμή. Πώς το επιλύεται αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, περιπτώσει για την προσπάθεια που καταβάλλατε διότι όλη η εργασία του κανονισμού, της οδηγίας είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα αλλάξουν άρδιν τα όσα συμβαίνουν και μία ερώτηση σχετικά με τις κυρώσεις. Στη χώρα μου αυτό δεν επαρκεί. Αυτές οι κυρώσεις δεν επαρκούν, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι ειδικευμένε στην συλλογή δεδομένων και τις κυρώσεις της πληρώνουν διότι κερδίζουν πολλά περισσότερα. Μόνο όλοι καταβάλουν και πρόστιμα. Εντάξει, μπορεί να τροποποιηθεί. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος από να λάβει το λόγο. Εγώ θα μιλήσω, θα θέσω την τελευταία ερώτηση. Έβαλα και το ρολόι να τρέχει. Ανησυχώ για το ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά μέσα, των οποίων το ένα, η οδηγία, παρουσιάζει πολύ χαμηλότερα επίπεδα προστασίας από ότι ο κανονισμός και στη δημόσια συζήτηση εστιάσαμε στον κανονισμό, λίγο στην οδηγία και νομίζω ότι αυτή είναι που παρουσιάζει ε, μεγαλύτερο κίνδυνο και διερωτώ με πώς η Κομισιόν επιλύει το ζήτημα όπου μια βάση δεδομένων που δημιουργηθεί για εμπορικούς σκοπούς χρησιμοποιείται για την επιβολή νόμου. Λοιπόν, ποια από τα δύο πρότυπα, ποια τα δύο στάνταρ εφαρμόζονται. Δεύτερον, εάν διαβάσετε τον τίτλο της οδηγίας, βλέπετε ότι υπάρχουν στόχοι που αλληλογροθοκοπούνται. Το ένα αφορά την προστασία ε, ε, θεμελιών δικαιωμάτων και το άλλο αφορά την ε, ποινικέ κυρώσει ε, και δίωξη αξιόμενων πράξεων. τι θα κάνει ο δικαστή, τι θα πει. Το άρθρο 16 που είναι η νομική βάση σαφώς αφορούν την, αφορά στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά μετά βρήκα ανησυχητικό ότι γίνεται διάκριση ανάμεσα σε ατομικές ε, περιστάσει και μαζικές ε, υποθέσεις και ένα άλλο στοιχείο είναι η μεταφορά δεδομένων σε τρίτα κράτη δίχως δικαστική επέμβαση. Δηλαδή εδώ ανοίγουμε την ε, πόρτα για μεταφορά δεδομένων σε άλλα κράτη δίχως να, να χρησιμοποιηθούν ή ε, να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι συνθήκες ε, αμοιβαίας συνδρομής. βλέπω ότι η Κομισιόν εδώ δεν προσπαθεί να προστατεύσει τις ήδη ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Παρακαλώ κυρία Γενική Διευθύντρια. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μία προς μία. Καταρχάς, κατεξουσιοδότηση πράξης. Κάποιοι από εσάς ανησυχήσατε για την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις, αυτές τις πράξεις της κατεξουσιοδότηση για να τροποποιήσει το 85% της σύμβασης. Κοιτάξτε, μια τέτοια πράξη κατεξουσιοδότηση δεν μπορεί να ανάξει το κανονισμό. Μπορεί να δώσει μια ερμηνεία ενός κανονισμού, και ε, ξαφνικά τώρα δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον κανονισμό. Οι προθέσεις μας είναι γνωστές, πρέπει να ακολουθήσουμε διαδικασίες μέσω επιτροπολογίας, μέσω κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν μια θεσμική διαδικασία. Δεν είστε οι μόνοι που ανησυχείτε για τις κατεξιοδότηση πράξεις, αλλά δεν είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αλλάξει επί της ουσίας ένα τέτοιο νομοθετικό, αν θέλετε, έγγραφο. Δεύτερο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γραφειοκρατική επιβάρυνση. Όπως σας είπα, προσπαθήσαμε να ελαφρύνουμε το βάρος για τις μικρομεσαίες. Γιατί? γιατί για τις περισσότερες μικρομεσαίες δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Και αν είστε μια μικρή ε, επιχείρηση με ένα κατάλογο πελατών και διευθύνσεων, Δεν χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, ειδικά μέτρα, δεν χρειάζεται ειδικό υπάλληλο υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κτλ. Πρέπει να διευκρινιστούν εδώ τα πράγματα. Δεν εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εφαρμογή του κανονισμού, μεν. Αλλά παρόλα αυτά το διοικητικό άχθος το οποίο συνδέεται με την εφαρμογή του κανονισμού είναι σαφώς ελαφρυμένο ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για το αν έχουμε ισορροπήσει τα πράγματα σωστά. Νομίζω ότι είμαστε δίκαιοι. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, για τη σύμφωνη γνώμη, τη συνένεση. Είναι σαφές ότι πρέπει να ότι η συνένεση είναι ένας, αν θέλετε, από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 6 υπάρχουν πολλές δυνατότητες νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων μέσω συμβάσεων προς το δημόσιο συμφέρον, θεμητών συμφερόντων κτλ. Όταν κάποιοι λέγουν λοιπόν ότι η συνένεση θα πρέπει να είναι η μοναδική βάση, το μοναδικό θεμέλιο, αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχουν έξι διαφορετικές διαδικασίες για νόμιμες νομικές επεξεργασίες δεδομένων. Όταν όμως απαιτείται η συνένεση και όταν επιλέξει ο επεξεργαστής ότι η συνένεση είναι προαπαιτούμενη, προφανώς η συνένεση αυτή θα πρέπει να είναι απολύτως εκπεφρασμένη. Σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει κανείς κάτι το οποίο να ξεκαθαρίζει ότι συμφωνεί μια δήλωση στο διαδίκτυο, κάτι εν Συνένεση μέσω αποχής <clears throat> δεν υπάρχει, μέσω αδράνειας δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει εκπεφρασμένη ε, βούληση. Συνδέεται με αυτό είναι το σβήσιμο κάποιων δεδομένων και το δικαίωμα του να ξεχαστούν κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε, εμείς δεν προτείνουμε ότι θέλουμε να γράψουμε ιστορία εμείς με την πρόταση αυτή. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ανασχεδιάσουμε την ιστορία και να την ξαναγράψουμε. Δεν ζητάμε εμείς αλλαγές ας πούμε για τους δημοσιογράφους και τα λοιπά. Αυτά θέλουμε να τα προστατεύσουμε, διότι η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι το θεμελιώδες και πρέπει να ισορροπήσουμε ε, το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των ιδιωτικών στοιχείων με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Και αυτό ακριβώς γίνεται στα πλαίσια της προτάσεώς μας. Τώρα θα αλλάξω γλώσσα, θα μιλήσω γαλλικά για την Γαλλίδα συνάδελφο, για τους λόγους τους οποίους ε, σας είπα κυρία Βερσά. Έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από άλλους. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Όχι, για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί οι βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη οδηγία είναι οι ίδιες με τις βασικές αρχές τις οποίες περιλαμβάνει ο κανονισμός. Για πρώτη φορά εμείς διευρύνουμε τις βασικές αρχές της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων στα πλαίσια της συγκεκριμένη οδηγίας και το κάνουμε όχι μόνο για την μεταφορά την διαμεθοριακή στοιχείων, αλλά το κάνουμε επίσης και για την εσωτερική διαδικασία, κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε. Αν θέλετε λοιπόν η βασική αρχή της οδηγίας δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε βασική αρχή είναι ότι από τη μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει προσφυγές επί παραλήψη, επί μάλλον, που δεν σέβονται τις ρυθμίσεις αυτές και αυτό είναι σημαντικό βήμα σε σχέση με τις αποφάσεις πλαίσιο που ισχύουν σήμερα. Θέσατε το ερώτημα επίσης το τι κάνουμε για τους ε, ευάλωτους πληθυσμούς. Αυτό το οποίο κάνουμε, παράδειγμα, είναι τα ειδικά μέτρα τα οποία παίρνουμε για τα παιδιά. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα άρθρο το οποίο διευκρινίζει ότι για τα παιδιά κάτω των 13 η συνένεση των γονέων είναι σαφής, είναι υποχρεωτική. Γι' αυτό εξετάσαμε πιο προσεκτικά αυτές τις κατηγορίες λοιπόν, τις πιο ευάλωτες του γενικού πληθυσμού. Τώρα οι διεθνείς συμφωνίες για τις διεθνείς συμφωνίες θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά δεν θα ήταν σωστό να το κάνω. Θα ήταν απρόσεκτο από πλευράς μου. Ο κανονισμός αυτός αφή στιγμής τεθεί σε ισχύ και η οδηγία τεθεί σε ισχύ κάποιες ειδικέ συμφωνίες όπως το PNR που περιλαμβάνουν αν θέλετε ρήτρε για προστασία δεδομένων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ε, τις δικές μας αυτές ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι αυτονόητο. Λέμε επίσης ότι δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση τις προϋπάρχουσες συμφωνίες, αλλά δεν τις αμφισβητούμε άμεσα, πολύ απλά, γιατί θα πρέπει να επαληθευτεί να ελεγχθεί αν οι ισχύουσες αυτές συμφωνίες βρίσκονται συμβατές με αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει ή με αυτά τα οποία θα αποφασίσουμε στο μέλλον στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων. Θέσατε και ένα ερώτημα για τις κυρώσεις. Και με ενδιαφέρει αυτό, γιατί οι αντιδράσεις τις οποίες είχαμε για τις κυρώσεις ήταν κάποιες, θα έλεγα, καταδικαστικές ουσιαστικά για μας αντιδράσεις, λέγοντάς μας ότι υπερβάλλουμε. Όχι. Καταρχάς προηγείται μια προειδοποίηση. Για αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται αυτά τα δεδομένα τους προειδοποιούμε ότι κοιτάξτε δεν τα σέβεστε, πάρτε τα μέτρα σας. Και μετά έρχονται οι κυρώσεις οι οποίες είναι διαφορετικού εύρους και μπορεί να είναι πρόστιμο που φτάνει μέχρι το 1 εκατομμύριο ή ένα σημαντικό ποσοστό του διεθνούς τζίρου των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό οι επιχειρήσεις ε, θα σκεφτούν πάρα πολύ προσεκτικά και αυτό είναι ο στόχος μας πριν πάρουν μέτρα τα οποία θα μας εκθέσουν θα τις εκθέσουν μάλλον σε ε, κυρώσεις τέτοιου βάρους που σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγνοήσει κανείς εύκολα. Και τώρα επιστρέφω στις δικές σας ερωτήσεις κύριε Εντεβέλτ που είναι πάντα για μένα οι πιο δύσκολες. Είπατε ότι είστε απογοητευμένοι γιατί δεν λύσαμε ακόμα το θέμα της μεταφοράς δεδομένων προς τρίτες χώρες. Και αυτό δεν γίνεται μέσω απόφασης δικαστικής. Πράγματι δεν περιλαμβάνεται η πρόταση αυτή ε, στη, δική μας νομοθετική πρόταση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να το διευκρινίσω αυτό. Υπάρχει αιτιολογική σκέψη 90, την οποία πρέπει κανείς να διαβάσει από κοινού με το άρθρο 24-7. Αυτό το οποίο λέγεται εκεί είναι ότι πιστεύουμε πως εάν μια εταιρεία, μια επιχείρηση της ζητηθεί από μια αστυνομική αρχή τρίτης χώρας να αποστείλει στοιχεία, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματα τουλάχιστον στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να περάσει μέσα από τα MRA είτε σε διμερές επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσφέρει ένα κάποιο επίπεδο προστασίας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε με τους Αμερικανούς φίλους μας. Και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε μία επιχείρηση στη δύσκολη θέση είτε να έχει να εφαρμόσει τον κανονισμό αυτό σε σχέση με τη συνεργασία με μια τρίτη χώρα είτε να παραβιάσει τον κανονισμό είτε του κράτους μέλους είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υπάρξει πρόοδος λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι διόλου εύκολο να ασχοληθεί κανείς μαζί του. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά εκ νέου Νομίζω ότι και στο Συμβούλιο γίνονται τα απαιτούμενα βήματα έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο ρυθμός των αλλαγών και θα θέλαμε και μαζί σας να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα από κοινού. Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε πολλές ανταλλαγές απόψεων τέτοιου τύπου στο μέλλον. και με ταχύτητα και με ομαλό τρόπο θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Η χρήση του PNR στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Κέρκοπφ. Thank you very much, Chairman. I really don't think we have enough time if we're going to finish on time here to do proper justice to this. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να κάνουμε μια κανονική συζήτηση. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αλλά όπως είπα δεν έχουμε αρκετό χρόνο και γι' αυτό οι σκιώδεις εισηγητές θα έρθουν σε επαφή μαζί μου όπως το ήδη το έχουν κάνει και θα θέσουν τις ανησυχίες τους και τα θέματα που τους απασχολούν. Υπάρχει και πολύ θόρυβο στην αίθουσα. Παρακαλώ ζητήστε από τους μη ενδιαφερμένους να αποχωρήσουν άμεσα. Παρακαλώ όσοι φύγετε να φύγετε χωρίς θόρυβο. Μην μιλάτε στους διαδρόμους. Λοιπόν χαίρομαι που έχουμε πια έστω και για λίγο την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της χρήσης του PNR στην Ευρώπη. Ελπίζω μέχρι τώρα όλοι να είχατε τη δυνατότητα να εξετάσετε τα δύο αυτά κείμενα. Το πρώτο είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το δεύτερο είναι η δική μου έκθεση, η οποία είναι μια απόκριση αν θέλετε στο κείμενο της Επιτροπής. Θα δείτε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαφοροποιούμε. Είχαμε ήδη μια μακρά συζήτηση για τα πιενά σήμερα και γι' αυτό δεν θα ήθελα να φανώ ιδιαιτέρως επαναληπτικός. Ελπίζω όμως ότι το κείμενο το οποίο σας έχω προτείνει να καλύπτει τις βασικές ανησυχίες τις οποίες έχετε εκφράσει εσείς σαν Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή όταν ξεκινήσαμε την εξέταση του θέματος. Στα πλαίσια της συγγραφής της νομοδότησής μου ήρθα σε επαφή και διαβουλεύτηκα και με τους καταναλωτές και με τις ε, αερομεταφορείς, με τις αστυνομικές και κατασταλτικές αρχές, με τις κυβερνήσεις και με τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους εμπλεκομένους στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είχαμε αρκετές συναντήσεις πληροφοριακές για το θέμα των δεδομένων PNR γενικά το οποίο είναι ένα από τα δύσκολα θέματα που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Να υπογραμμίσω συνοπτικά τα βασικά προβλήματα όπως τα βλέπω, θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε. Πρώτον, το εάν το θέμα αυτό είναι ένα ενδοκινοτικό θέμα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη και υπάρχει προστιθέμενη αξία για ένα σύστημα το οποίο να μην αφορά μόνο τις πτήσεις από τρίτες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό των πτήσεων των, χωρών. Υπάρχουν εκατομμύρια πτήσεις οι οποίες ε, περνούν από την Ευρώπη, έχουν σταθμούς στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα σημαντικό θέμα γύρω από τις δραστηριότητες των τρομοκρατών και των ε, ε, εγκληματιών οι οποίοι σκοπεύουν να διαπράξουν τέτοιες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιλέγουν βέβαια τον ευκολότερο δρόμο, δεν συμπεριφέρονται όπως οι κανονικοί άνθρωποι, πολλές φορές σβήνουν τα ίχνη τους και είναι δύσκολο να τους παρακολουθήσει κανείς. Υπάρχουν εκατοντάδες δρόμοι για να φτάσει κανείς στην Ευρώπη σήμερα. και μη παρακολουθώντας τις εσωτερικές πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουμε τη δυνατότητα στους εγκληματίες να διευκολύνουν την προετοιμασία των εγκληματικών τους ενεργειών. Δεύτερον, να αναφερθώ τώρα στο θέμα της προστασίας των δεδομένων των προσωπικών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια των εμπειριών που έχουμε συλλέξει, στα πλαίσια των συμφωνιών PNR και άλλων, να πω ότι η συγκεκριμένη αυτή συμφωνία δεν θα πρέπει να ταυτιστεί με τις υπόλοιπες, διότι υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι, βλέποντας το τι πραγματικά είναι. Δεν είναι μία διαπραγμάτευση με μία τρίτη χώρα, δεν είναι μία διαπραγμάτευση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι το οποίο αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προστασία της. Έκανα πολλές αναφορές στην έκθεσή μου και στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στα άρθρα 8 και 21. Οι περισσότερες αλλαγές και προσθήκες στο κείμενο της Επιτροπής, τις οποίες προτείνω εγώ, αφορούν την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Λέγεται στην πρόταση ότι οι επιβάτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να ελέγξουν να ζητήσουν αποζημίωση και δικαστική αποκατάσταση όπου αυτό χρήζεται απαραίτητο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λάβουν δράση εναντίον αυτών οι οποίοι στρεβλά χρησιμοποιούν μέσω της λειτουργίας του συστήματος τα προσωπικά δεδομένα όπως άρνηση ε, χρήσης του συστήματος, μομφή και πολλές φορές να περάσουν και στην απαλλαγή από τα καθήκοντα των αξιωματικών οι οποίοι έχουν παραβιάσει τις ρυθμίσεις. Ανάλογα με τον κώδικα συμπεριφοράς, η επεξεργασία των δεδομένων PNR και αυτοί οι οποίοι κάνουν την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να είναι στόχος αυστηρής και ε, συγκεκριμένης διαδικασίας κατάρτισης και θα πρέπει να περιορίζονται στο να, σε σχέση με τα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Και θα πρέπει επίσης να δούμε εδώ και τη δυνατότητα δημιουργίας εθνικών αρχών οι οποίες να ελέγχουν τις διαδικασίες αυτές και να υπάρχει και μία περίοδος ελέγχου αξιολόγησης και αναθεώρησης πιθανώς, προτείνω την πενταετία, και να σας διευκρινίσω λίγο και αυτό το οποίο ονομάζω masking out, δηλαδή απόκρυψη δεδομένων εκ των υστέρων. Υπάρχει τώρα και το θέμα της συγκράτησης των στοιχείων, της διάρκειας συγκράτησης τους. Τα στοιχεία PNR, τα οποία μας δίδουν οι αερομεταφορείς στη μονάδα πληροφοριών επιβατών, θα μένουν εκεί για 30 μέρες μετά από την μεταφορά τους στη συγκεκριμένη υπηρεσία από την χώρα στην οποία πήγε, την πρώτη χώρα στην οποία πήγε ο επιβάτης. Μετά η ε, συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να κρατήσει τα στοιχεία αυτά για μια περαιτέρω περίοδο πενταετή. Αυτό είναι κάτι με το οποίο έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ελπίζω να βρεθεί εκ νέου μια κάποια συμφωνία. Και τώρα ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος. Εδώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και των κρατών μελών και των υπηρεσιών τήρησης τάξης ε, είναι θα έλεγα κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί για να λειτουργήσει το σύστημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν μυστικά για τα επιτυχή και μη επιτυχή χαρακτηριστικά του συστήματος και θα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η συγκεκριμένη πρόταση. Η Επιτροπή ως θεματοφύλακτη συνθήκης μπορεί να κάνει μια τεχνική αξιολόγηση του συστήματος έτσι ώστε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των επιβατών και το Κοινοβούλιο να μπορεί να είναι σε θέση ξεκάθαρα να δει αν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το σύστημα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως βλέπετε από την έκθεση λέγεται ότι θα υπάρχει ένα πολυστρωματικό θα έλεγα σύστημα ελέγχων. Οι δράσεις συστηματικά θα ελέγχονται, θα αξιολογούνται και τώρα σχετικά με το κόστος. Όταν βλέπει κανείς το μέγεθος των δαπανών των κρατών μελών στην τήρηση της τάξης και στην άμυνα γενικότερα, βλέπουμε ότι το κόστος που απαιτείται εδώ είναι κάτι το πάρα πολύ λογικό για την προστασία των χωρών και των πολιτών της Ένωσης. We that the Προτείνουμε η περίοδος για τον, που θα απαιτηθεί για τον καθορισμό στα κράτη-μέλη να ξεκινήσει στα τρία χρόνια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν το σύστημά τους με σωστό τρόπο και τεχνικά και οικονομικά. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο ε, συνομιλούντες με τους εκπροσώπους των αερομεταφορέων. Θα πρέπει οι επιβάτες να έχουν επιλογές με βασική και πρώτη επιλογή την ασφάλειά τους. Μας διασφαλίστηκε ότι το κόστος για τον επιβάτη δεν θα ξεπεράσει κάποια ε, θα έλεγα εκατοστά ευρώ ουσιαστικά ανά ε, ε, εισιτήριο. Νομίζω ότι το τίμημα είναι πάρα πολύ χαμηλό γιατί μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη εγκληματιών και είναι τίποτα αμεληταίο σε σχέση με επιπλέον κόστη των αερομεταφορών όπως το κόστος μεταφοράς αποσκευών, διαχείρισης εισιτηρίων κτλ. Τώρα, η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα. Τα συζητήσαμε σήμερα αυτά και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε σε σχέση με τέτοιου είδους θέματα. Εγώ για πάρα πολύ καιρό πίστευα ότι η οδηγία αυτή είναι απαραίτητη. Νομίζω ότι είναι ένα αξιόλογο μέσο στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Είναι μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, να συνεργαστούν καλά στην ανταλλαγή δεδομένων σε ένα πλαίσιο το οποίο να διευκρινίζει τα νομικά όρια και να είναι χρήσιμο και για τον επιβάτη και για τον αερομεταφορέα. Στα πλαίσια αυτού του πολλαπλού συστήματος ελέγχου και σεβασμού των κανόνων στο οποίο προαναφέρθηκα. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα συντονισμένο σύστημα με συγκεκριμένους κανόνες ελέγχου. Τα δεδομένα PNR είναι πληροφορίες τις οποίες εμπιστευόμεθα και στέλνουμε και στους συμμάχους μας σε τρίτες χώρες. Τουλάχιστον ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό λοιπόν με κάποιους συμμάχους ε, και τρίτες χώρες, τότε μπορούμε να το κάνουμε φυσικά και μεταξύ μας. Έχουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη που απαιτείται. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία είναι μια η δυνατότητα για να δημιουργηθεί ένα μέσο ασφάλειας συμβατό με τις ευρωπαϊκές αξίες και η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι το οποίο όλοι υποστηρίζουμε. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου, Πρόεδρε. Δεν θέλω να περάσω σε όλες τις τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει γιατί τις έχετε μπροστά σας, αλλά θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και εγώ θα συζητήσω τα θέματα αυτά συνολικά με τους σκιώδεις εισηγητές και θα ακούσω με χαρά τις απόψεις τους. Δεν είμαστε και πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Τέσσερις. Πέντε. Λοιπόν, το λόγο έχουν ε, τα μέλη και θα ακολουθήσει η Κομισιόν και το Συμβούλιο για να απαντήσουν σύντομα. Ο κύριος Βος, ε, να ζητήσω από όλους σας ε, να είστε λακωνικοί. 1,5 λεπτό έκαστος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή. Έκανε πολύ καλή δουλειά και πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ για τα συμπληρωματικά της ε, δουλειάς του που μας καθοδηγούν. Θα ήθελα να πω ότι κατά βάση θα πρέπει, εφόσον περάσει το PNR, να έχουμε και τα συνοδευτικές προτάσεις του κυρίου Κύρκοπ. Επτά κέρια σημεία, μάλλον τέσσερα, δύο αρνητικά, δύο θετικά. Δύο αρνητικά δεν διαφαίνονται πλοίο ψηφίες, πράγμα το οποίο Ίσως θα εξασφαλίζονταν αν είχαμε μείνει στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον χώρο του Σέγγεν, θα μπορούσαμε να περιμένουμε έναν ασφαλή χώρο και ανάλυση δεδομένων με όχι τόσο υψηλό βαθμό προτεραιότητας, δηλαδή να είχαμε εξασφαλίσει διαφορετικά την ασφάλεια. Επίσης η ελευθερία της ε, κυκλοφορίας των πολιτών, της εκκίνησης στο πλαίσιο του χώρου του Σέγγεν, ε, δεν επιτρέψει σε κανένα να παρεμποδίσει το δικαίωμα να ταξιδεύει. Οι προπολογισμοί για το PNR, για άλλη μια φορά θα φέρω το θέμα αυτό, πρέπει να έχουμε στο δυνατόν καλύτερη λύση, οικονομική λύση βέβαια, αλλά και αποτελεσματική λύση στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα είμαστε στο δυνατόν πιο σύντομος πρόεδρε, Θεωρώ λοιπόν ότι ο χρόνος ε, της διακράτησης των δεδομένων, η ανάλυση του κινδύνου, η μέθοδος διαβίβασης ε, στα τρίτα κράτη, οι όροι, ε, η διαφύλαξη των, ασφαλ... των ευαίσθητων δεδομένων και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικέ διαστάσεις. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος και λυπούμε τους διερμηνείς, ο κύριος Άλμπρικτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση της έκθεσης τον κύριο Κέρκοπ. Όντως είναι καλή συνεργασία μαζί του και έτσι στο θέμα αυτό διαφοροποιούμαστε σημαντικά ως προς το πόσο είναι απαραίτητο και αναγκαίο το πλαίσιο τέτοιων μέτρων όπως αυτά προτείνατε. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Κόστος το οποίο θεωρώ άλλωστε ακούστηκε και νωρίτερα σημαντικά υψηλότερο από ό,τι είχαμε αρχικά ακούσει. Θα κοστίσει το σύστημα αυτό και λόγω των πληροφοριών, του αριθμού, του όγκου των πληροφοριών που συλλέγονται, βάσει των όσων προβλέπει τουλάχιστον η έκθεση, ε, το σχέδιο εκθέσεως, θα είναι σχετικά υψηλό για τις ε, αεροπορικές εταιρείες. Και επιπλέον Δεύτερο σημείο. Εάν αρχίσουμε να καταγράφουμε όχι μόνο τις ε, διεθνείς, δηλαδή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση πτήσεις, αλλά και τις εσωτερικές, τότε αυτό θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες. Επιπλέον δε η, διάσταση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων παραμένει. Η α, επικρίσεις που διατυπώσαν ως προς την PNR για τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν και με την ίδια έμφαση και ένταση διατυπώνονται και σε αυτήν την περίπτωση. Ευχαριστώ, η Βαρόνι Λάτφορντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με παραξενεύει η διευκρίνηση του Τίμωθη ως προς το ανομιμοποίηση και κάλυψη, Anonymize και masking out. Ε, και σε σύγκριση για την με την πρόταση Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η διαφορά, διότι εγώ νόμιζα ότι οι πληροφορίες ήταν απόκριφες, ε, συγκαλυμμένες δηλαδή και ανώνυμες ήδη, masked και anonymized. Άρα με τη διαφοροποίηση που κάνει ο κύριος Κέρκοπ με προβληματίζει στην τροπολογία 22 που αναφέρεται στο masking, ως όχι απαραίτητα απάλληψη του ονόματος του επιβάτου, πράγμα το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ε, ωστόσο, η ερώτησή μου για τις ιστορικές τετραπτήσεις έχει να κάνει με το εξής. Ε, καταλαβαίνω αυτό που λέει για τις ε, ανταποκρίσεις, αλλά γιατί πρέπει να συνεργάζονται οι αρχές των κατώμερων. Εντάξει, να καταλάβω ότι αν υπάρχει δυνατότητα ε, για τους... Ε, ή αν θεωρούν οι ε, λαθρέμποροι ναρκωτικών ότι μπορούν να αντιπαρέλθουν τον κίνδυνο του ελέγχου από τις αρχές μέσω μιας διαφορετικής, ενός διαφορετικού δρομολογίου, δεν θα χρειάζεται ούτως ή άλλως συνεργασία μεταξύ των κρατών. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ουσιαστική συνεργασία μας μεταξύ των αρχών και όχι όλο και πιο, πολλές, πιο πολλά στοιχεία που συλλέγονται. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. ευχαριστώ τον κύριο Κίρκοπ για την προσπάθεια που κατέβαλε. Γεγονός είναι ότι εγώ έχω επί της ουσίας προβλήματα με την έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα διότι αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία αφορά μια νέα τεχνολογία αυτή της, του περιορισμού της συλλογή. Ε, το, το πρόγραμμα δεν αναφέρεται το ευρωπαϊκό έλλειμμα που έχουμε, αλλά αναφερόμαστε στο ευρωπαϊκό PNR. Γιατί κατεπήγον το θέμα. Είναι γεγονό ότι η δικαστική και αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη βρίσκεται στα ελάχιστα επίπεδα. Τα ακούγαμε σήμερα και με την παρουσία της Europol και το τι κάνει η Ευρώπη με το TFTP. Αυτή λοιπόν η συνεργασία η οποία βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, ακόμα και μέσα στην Ευρώπη, το πλαίσιο για το οποίο μιλάμε εδώ είναι κάτι το καινούριο, μια νέα φιλοσοφία που αφορά αυτήν την αστυνομική δικαστική συνεργασία. Ήδη δεν βελτιώνουμε αυτήν τη συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να αιτιολογήσουμε το κατεπήγον οι εμπειρογνώμονε γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό το μέσο δεν αφορά το, και το μέτρο δεν αφορά την τρομοκρατία και αν δεν αφορά την τρομοκρατία αλλά ούτε την, ε, το οργανωμένο έγκλημα, κάτι το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρώ ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Πολλά απομένουν να γίνουν. Δεν μπορώ να εκφράσω άλλα επιχειρήματα διότι υπάρχουν πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Τρία θέματα, Πρόεδρε. Το πρώτο αφορά στο κόστος. Οι αστυνομικές αρχές μου είπαν και μπορεί να έχουν άγνοια, αλλά πρέπει να τους δυσπιστήσουμε ε, μέχρι τώρα. Ότι αν το Λουξεμβούργο πρόκειται να εφαρμόσει ένα τέτοιο σύστημα, θα αντιμετώπιζε ένα κόστος 30 50 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι αμεληταίο ποσό, αλλά πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει σχέση με το γεγονό ότι έχουμε ένα και μόνο αεροδρόμιο στη χώρα μου και ότι θα συμπεριλάβουμε ε, πτήσεις ενδοευρωπαϊκές ε, νομίζω ότι αυτό θα ε, είναι ένα μέτρο περιορισμού της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά Τώρα, για την έννοια του σοβαρού εγκλήματος μπορεί να θεωρηθεί κάτι το οποίο οδηγεί σε, μια, ε, σε φυλάκιση τριών ετών. Μα κοιτάξτε, στη δική μου τη χώρα κάποιος που κλέβει ποδήλατο για τρία χρόνια καταδικάζεται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί απειλή για την ασφάλεια, ούτε για την προσωπική μου, ούτε για την εθνική. Και τέλος, ο εισηγητής ε, ενδεχόμενα έχει δίκιο όταν ε, λέει ότι οι οδοί της ε, τρομοκρατίας έχουν καταστεί δύσκολα ε, δεν μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα, δύσκολα, εύκολα συγγνώμη. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ το πρόβλημα αφορά ιδιαίτερα τις αεροπορικές εταιρείε χαμηλού κόστους ε, κοιτάξτε, καλύτερα να ταξιδεύουμε με ποδήλατο παρατηρεί ο πρόεδρος. Ε, ε, Ματιού, να συγχαρώ τον κύριο Κίρκοπφ. Πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα τη συμφωνίας με τρίτες χώρες. Εγώ θα ήθελα μια πλήρη πρόσβαση στα PNR για μια περίοδο ενός έτους, διότι η εμπειρία δείχνει ότι οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες κάνουν πολλαπλά ταξίδια εντός ε, Ένωσης ε, και μεταβαίνουν στις χώρες ε, στόχο των δράσεών τους. Λοιπόν, όταν έχουμε συγκαλυμμένα δεδομένα, δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. λοιπόν θα πρέπει η διάρκεια να είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι πρόσβαση στο PNR από την προλεπόμενη. Ευχαριστώ. Να πω κάτι. Είδα ότι κάποιες προτάσεις του εισηγητή βελτιώνουν την πρόταση της Κομισιόν, αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα που με ανησυχούν. Το ένα είναι οι ενδοενωσιακές πτήσεις. Ίσως πρόκειται για παραβίαση των κανόνων Σέγγεν, ε, διότι μιλάει για ελέγχους στα σύνορα και το ζήτημα επίσης ε, των μεταφορών. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, να το ξέρουμε πολύ προσεκτικά, γιατί δεν υπάρχουν ε, οι κατάλληλες προβλέψεις περί προστασίας. Και Σπίμπη είναι εδώ. Ευχαριστώ. Ο χρόνος τρέχει. Χαίρομαι που ξεκινήσατε να δουλεύετε επί της προτάσεως. Το Συμβούλιο προχωράει γρήγορα. Κάποια σημεία που εθίγησαν σήμερα το απόγευμα και ελπίζω θα έχουμε κάποια άλλη ευκαιρία να μπούμε σε λεπτομέρειες ε, όπως γνωρίζετε η ε, Κομισιόν σε αυτό το στάδιο αποφάσισε να προτείνει μια προοδευτική βήμα προς βήμα εξέταση, μάλλον πρόταση. Δεν έχουμε ακόμα συμπεριλάβει τα ενδοενωσ... τις ενδοενωσιακές πτήσεις. Θα είπα ότι θα κάνουμε αυτή την προσέγγιση βήμα προς βήμα, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι σοφρονέστερο έχοντας κατά νου ότι τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνει το σύστημα PNR για τις ε, ενδοκοινωτικές ε, πτήσεις ε, και το κόστος είναι κάτι το οποίο μας καθοδηγεί. Τώρα για το κόστος είναι σοβαρό ζήτημα συζητήσεις που έχουμε με τα κρατημέλη και στο για το Συμβούλιο. Σίγουρα αυτά τα προγράμματα κοστίζουν. Είχαμε μακροσκύλες συζητήσεις και με το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας ε, σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Υπάρχει δυνατότητα ε, συνδρομής ε, της Ευρωπαϊκή Ένωσης προς τα κράτη-μέλη. Όντω το κόστος είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν θελήσαμε ε, εξ αρχής να συμπεριλάβουμε τις ενδονοσιακές πτήσεις στην πρόταση. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλές από τις τροπολογίες ε, του εισηγητή. Θα μπορούσα να σας αναφέρω 25 αριθμούς, αλλά εμπεστώσει υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, που χρειάζεται να τις εξετάσουμε λίγο παραπάνω. Το θέμα του μοιράσματος των ε, δεδομένων με άλλα κράτη-μέλη, το θέμα της ε, privacy, Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν καλύπτονται από τις προτινόμενες τροπολογίες. Θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω την διατύπωση. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Όντως κατέβαλε σημαντική προσπάθεια. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής ε, θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Α, συγγνώμη. Ξέχασα τη Δανική Προεδρία. Σύντομα παρακαλώ. Έχουμε έξι λεπτά γιατί οι διερμηνείς μας έδωσαν 10 συνολικά λεπτά από τον χρόνο τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Το Συμβούλιο Χρειάζεται λίγο χρόνο να εξετάσει πιο αναλυτικά το έγγραφο. Νομίζουμε όμως ε, ότι σε πολλά συμφωνούμε. Χαιρόμαστε που το γεγονός ότι ο Ιζήτης έχει συμπεριλάβει και στο πεδίο εφαρμογής ε, τις ε, ενδοενωσιακές πτήσεις ε, ακόμα δεν έχει αποκρισταλωθεί άποψη στο Συμβούλιο αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφώνησαν ε, σε εθελούσια βάση για τη συμπερίληψη των, ενδο, πτήσεων. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση και του σοβαρού εγκλήματος. Να πω επίσης ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την οδηγία PNR ε, Ήρθαμε σε επαφή με τις εμπλεκόμενες αρχές ε, των κρατών μελών, οι οποίες ε, μας έδωσαν στοιχεία για την χρήση του PNR για θέματα διαρεύνησης και διαπίστωσης σε περιπτώσεις σοβαρού εγκλήματος και ότι πολλές αρχές θεωρούν ότι η χρήση του PNR είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή εργασία τους και θα ήθελα να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο για την διαχείριση αυτών των δεδομένων. Ορισμένοι βουλευτές μίλησαν για το κόστος και ο κ. Σπρίβ επίσης αναφίβολα είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και για το Συμβούλιο, όπως ε, φαντάζεστε. Γίνανε συζητήσει σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε συζήτηση στο άτυπο Συμβούλιο τον Ιανουάριο, όπου αποφασίστηκε πως ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε ένα μελλοντικό κανονισμό ε, σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριος Κίρκοπφ. Μισό λεπτό έχω. Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις όπως θα ήθελα πληρώς. Ε, απλώς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σημείωσα πολύ προσεκτικά τα όσα είναι συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσει και με τους σκιώδης συγκητές. Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση τα πρόκειται για εσωτερικίες ή μη ε, κινήσεις. Εάν θα περιλάβουμε και τις εσωτερικές θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αργότερα, γιατί μου φαίνεται λίγο προγραμματικό. Για την σταδιακή εισαγωγή έχω μια μάλλον αρνητική εμπειρία. Αναγκαιότητα, ο κύριος Άλπρεχτ βεβαίω έχει δίκιο να ρωτάει εάν είναι αναγκαίο να εισαχθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο και για την τροπολογία της ε, κυρίας Λάτσφορτ μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο το masking out διμερός. Για δε το κόστος θα καλυφθεί πιστεύω. Το σημείο του κόστους, το θέμα του κόστου είναι σημαντικό και πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω και εγώ πρέπει να βεβαιωθώ για το ποιος θα ε, έχει την επιβάρυνση αυτή με αυτή τη δαπάνη. Πάντως δεν βιάζομαι να προχωρήσει αυτή η πρόταση γρήγορα, βιάζομαι να προχωρήσει σωστά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και επειδή άκουσα βέβαια τους συναδέλφους, αλλά και επειδή είμαι πάντα ανοιχτό σε προτάσεις, υποδείξεις που ενδεχομένω προηγούνται από συνεδριάσεις ε, ε συγητές, θα περίμενα με πολύ μεγάλη δημονία μια περαιτέρω συζήτηση στο θέμα αυτό και ευχαριστώ βέβαια και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο, η Πρόεδρος. Μου θυμίζει αυτή η παρατήρηση για, το, για, τη, για σταδιακή εισαγωγή, την ε, σταδιακή εισαγωγή της οδήγησης στα αριστερά στην, ε, των δρόμων. 12 Μαρτίου το μεσημέρι, αν δεν κάνω πρόεδρε, είναι η κατάθεση για την, ε, η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Καλώς. Ευχαριστούμε τους Ερμήνες, λέει η Πρόεδρος. Χαίρετε.